Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να αρχίσουμε σιγά σιγά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και να μπούμε αμέσω στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα τα διαδικαστικά. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, αν δεν διαφωνεί κανείς, θεωρείται εγκεκριμένη η ημερήσια διάταξη. Προχωρούμε αμέσως στο σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα να σας ε, πληροφορήσω και πάλι ότι ε, μεταδίδεται απευθείας ε, στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και έχουμε διερμηνία σε 20 από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, μπορούμε να περάσουμε αμέσως στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Πολλών συνεδριάσεων, 25-26 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου, 7 και 8 Οκτωβρίου. Και αν δεν διαφωνεί κανείς, θεωρούνται εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Και θα περάσουμε αμέσως στο σημείο 4 τώρα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα, σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστοσης για τις εισαγωγές βοήου κρέατος υψηλής ποιότητας. Η συγητής μας είναι ο Χέρμπερτ Ντόρφμαν. Θέλει το λόγο ο συντάκτης νομοδότησης. Σύντομα. Όχι, όχι. Μπορούμε να περάσουμε αμέσως στην ψηφοφορία. Θαυμάσια. Μπορούμε λοιπόν, χωρίς περαιτέρω συζητήσεις, να περάσουμε αμέσω στην ψηφοφορία. Δεν έχουμε ονομαστικές ψηφοφορίες. Υπάρχει μια τροπολογία μόνο. Απλή ψηφοφορία θα κάνουμε για την τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. So, dann brauchen wir Τώρα θα πρέπει να κάνουμε και την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έχετε Όλη τις κάρτες σας. Υπάρχει κανείς που να την ξέχασε. Όχι. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. So, dann schließe ich die Abstimmung. Πέρας εγκρίνεται η έκθεση. 33 υπέρ, 7 κατά. Συγχαρητήρια. Θερμά. Προχωρούμε. Στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Είναι αντίστοιχο το θέμα, αλλά αυτή τη φορά έχει να κάνει με την Ουκρανία. Συντάκτης ρομοδότησης είναι ο συνάδελφος Κούσμιουκ. Δεν ξέρω θέλει ξανά το λόγο. Όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω. Ωραία. Μπορούμε και εδώ να περάσουμε αμέσω στην ε, ψηφοφορία. Εδώ έχουμε δύο τροπολογίες. Okay. Änderungsantrag. Ε, είναι η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. Η τροπολογία παριθμό 2 ε, ψηφίπε, Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά και μπορούμε να περάσουμε και εδώ στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. και τελειώνει. «34 υπέρ, 9 κατά». Με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Και τελειώσαμε ήδη τις ε, ψηφοφορίες μας και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπαρίθμ 6 παρουσίαση των εργασιών του θεματικού τμήματος για τις διαρθρωτικές πολιτικές και την πολιτική συνοχής. Θα πρότεινα να το συζητήσουμε μαζί με το 7, δηλαδή να ακούσουμε πρώτα τις δύο παρουσιάσεις και μετά ε, να ε, ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις των συναδέλφων. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, στην Επιτροπή μας ε, τον κύριο Λίτσελμαν και του δίνω μέσω στο λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά που έχω την ευκαιρία σύντομα να σας παρουσιάσω το ρόλο του Τμήματος Πολιτικής και να ξεκινήσω τη σημερινή παρουσίαση στην αρχή αυτής της νέας κοινοβουλευτικής θητείας. Η το Τμήμα Πολιτική δημιουργήθηκε το 2004 για να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τη δουλειά των Επιτροπών στον τομέα τη έρευνα και τη εμπειρογνωμοσύνη. Όλε οι επιτροπέ του Κοινοβουλίου υποστηρίζονται από ένα τέτοιο τμήμα πολιτική, όπω δείχνει και αυτή η διαφάνεια. Το δικό μα τμήμα πολιτική, τέλο πάντων το δικό σα, το B, για την ε, διευθυντική πολιτική και την πολιτική συνοχή, έχει να κάνει με την DG Trade, Red, Envy και τη δική σα. Όπως είπα, παρέχουμε μελέτες ερεύνας σε κοινοβουλευτικά όργανα, όχι σε επιμέρους μεμονωμένους βουλευτές. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμάστε, καθώς αυτή είναι βασική διάκριση μεταξύ του δικού μας τμήματος πολιτικής και των, ε, του EPRS, του Τμήματος Μελετών για τα μέλη και το οποίο συντάσσει απαντήσεις στις δικές σας μεμονωμένες ερωτήσεις. Η εμπειρογνωμοσύνη που παρέχουμε χαρακτηρίζεται από την επικέντρωσή μας στην δράση. Θέλουμε να επικεντρωνόμαστε σε υποθέσεις πολιτικής και σενάρια τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη δικασία λήψη αποφάσεων για σας καθημερινά. Θέλουμε δηλαδή να διευκρινίσουμε νομικές, οικονομικές ή τεχνικές ε, διοργανωτικές πτυχές ή να δούμε τη μεταφορά και υλοποίηση της νομοθεσίας καθώς και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στόχος είναι να παρέχουμε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη για να μπορείτε και εσείς να προγραμματίσετε εγκαίρως τις στρατηγικές σας προτεραιότητες. Αυτό είναι καθοριστική σημασία, ώστε να μην, γίνουμε αυτό που κάνουμε, να μην γίνει αυτό που κάνουμε, να μην γίνει μια άσκηση ως αυτός σκοπός, ε, και τη θεωρητική μελέτη, αλλά να επηρεάσει την καθημερινή σα δουλειά. Επικεντρωνόμαστε στα διαφανή, αντικειμενικά και ανεξάρτητα στοιχεία και αυτό το επιδιώκουμε μέσα από διαγωνισμούς τους οποίους διαφημίζουμε και μάλιστα δραστηρία. Έχουμε πολύ αυστηρούς όρου και προποθέσει και επιλέγουμε του συμβαλωμένου με αυστηρή διαδικασία η οποία διοργανώνεται από δημοσίου υπαλλήλου που δεσμεύονται από το εσωτερικό κατανομισμό για τους υπαλλήλου και την ε, διοντολογική προσέγγιση. Βεβαίω έχουμε και μελέτες ομοτήμων και χρησιμοποιούμε ε, εργαλεία αξιολόγηση και βεβαίως το τελική δοκιμή είναι αυτή που περνάμε από εσά εδώ στην Επιτροπή σα, για να δούμε αν μα θεωρείτε και χρήσιμου. Τώρα, τα διάφορα είδη εμπειρογνωμοσύνη. Έχουμε τα σύντομα σημειώματα, τα σημειώματα τα ενημερωτικά, αλλά βασικά οι μελέτε των 36 σελίδων, όπω η σημερινή είναι το βασικό μα έργο. Θα πρέπει σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρω ότι όλες μας οι μελέτες συντάσσονται και δημοσιεύονται μόνον στα αγγλικά. Αυτό λόγω των περιορισμών που έχουμε σε ό,τι αφορά τις μεταφραστικές υπηρεσίες και την έμφαση που δίνουν αυτές στις εκθέσεις και τις τροπολογίες καταρχάς και μετά σε όλα τα άλλα. Προσπαθούμε τις γλωσσικές μας υπηρεσίες να τις ε, επεκτείνουμε όσο γίνεται και αυτό θα το δείτε και ε, στην επόμενη μελέτη όπου η με υπερίληψη, το executive summary έχει μεταφραστεί στις έξι βασικές γλώσσες εργασίας της Επιτροπής. Τώρα, εμπειρογνωμοσύνη που σας παρέχουμε, είτε από τους συνεργάτες μας in-house εδώ στο Κοινοβούλιο μπορεί να παραχθεί, είτε εκτός. Βεβαίως, έχουμε μόνο δύο υπαλλήλου που εργάζονται στο δικό σας τομέα, ο κ. Αρμπέρ Μαχσό και ο κ. Φεσουά Νέγκ. Δεν έχουμε πάρα πολλές ε, δυνατότητες. Το 95% λοιπόν των μελετών μας παραγγέλλονται εξωτερικώς. Είναι το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών, των διαγωνισμών που σας ανέφερα και χρησιμοποιούμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι διαδικασίες είναι τύπου δημοσίων προμηθειών και έχουν έτσι δομιονέκτημα τη χρονική προθεσμία. Χρειάζεται πολλή χρόνο για να ετοιμαστούν οι μελέτε που έχετε παραγγείλει. Και όπω δείχνει και η διαφάνεια, όλα ξεκινάνε με τις αποφάσεις των συντονιστών σας για μια συγκεκριμένη μελέτη. Μετά χρειάζονται έξι εβδομάδες έως τέσσερις μήνες για τη διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού και μετά δύο ως έξι μήνες ώστε ο συμπελόμενος να συντάξει, να συντάξει τη μελέτη και μετά ένα ως δύο μήνες για να ετοιμαστούν όλα να μεταφραστούν και τελικά φτάνουμε ένα χρόνο σχεδόν από τη στιγμή που παραγγέλλεται από την Επιτροπή σα και φτάνει να παρουσιαστεί εδώ. Τέσσερι, τεσσερισήμιση μήνε έω ένα χρόνο. Πρέπει λοιπόν να έχετε αυτό το χρονικό όριο ε, στο νου σα όταν θέλετε να συνδυάσετε μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία με μια μελέτη. Επί παραδείγματο. Βεβαίω, όλα τα κείμενά μα είναι δημοσιοποιημένα, έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτε στο διαδίκτυο και στο intranet DG Υπάρχει και το site της Επιτροπής. Έχουμε το δικό μας blog για τις έρευνες της Επιτροπής. Έχουμε Twitter. Και βεβαίω μπορείτε να τα βρείτε ατυπωμένα και στη βιβλιοθήκη. Ή αν μας ε, γράψετε να σας τα στείλουμε σε Άρτημα. Πολύ σύντομα ήθελα να σας πω τι έχουμε ετοιμάσει για την Επιτροπή Άγκρη στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και τι ετοιμάζεται τώρα. Τι βρίσκεται υπό εξέλιξη δηλαδή. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική φοιτεία είχαμε 39 εξωτερικές μελέτες, όπως βλέπετε, με μια, με μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως κίνδυνοι και ευκαιρίες για τον τομέα παραγωγής τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ενδεχόμενη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, τη σύγκριση των εισοδημάτων των γεωργών και κτηνοτρόφων στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις επιπτώσεις της κλιματικής πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γεωργία. Επίσης, για τις διευθυντικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, τις επιπτώσεις του Brexit, αλλά και εσωτερικές μελέτες που συντάξαμε, όπως την σύγκριση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και σε σχέση με το τι ισχύει τώρα κανονισμούς. Οι δύο μελέτες που ετοιμάζουμε τώρα για φέτος, θα τα δείτε σε δύο λεπτά, είναι οι μεγάλες τάσει στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, ε, παγκόσμια επισκόπηση και ενδεχόμενες πολιτικές απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Προοπτική και μετά η απασχόληση στον χώρο της Γεωργίας, οι τωρινές προκλήσεις και οι μελλοντικέ προοπτικές. Σε ό,τι αφορά το ερχόμενο εξάμεινο για το 2020, Θα συζητήσουμε με τους πολιτικούς συμβούλους για να δούμε τι ιδέες υπάρχουν για μελλοντικές μελέτες. Η πρόταση αυτή μετά θα υποβληθεί στους συντονιστές, προκειμένου να την σκεφτούν και να την εγκρίνουν. Και να πω ότι είναι προς όφελός μα να χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό και το κονδύλιο για τις μελέτες αποτελεσματικά και αυστηρά για να υπάρχει υποστηθέμενη αξία για τη δουλειά σα. Γι' αυτό λοιπόν σα καλώ πραγματικά να μα στέλνετε τι αντιδράσει σα και τι συμβολέ σα για, ε, για τον προγραμματισμό των μελλοντικών μελετών. Για να είμαστε βεβαίοι ότι αυτό που σα στέλνουμε είναι αυτό που ακριβώ χρειάζεστε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ja, Ευχαριστούμε κύριε Λίτσελμαν για αυτή την παρουσίαση. Νομίζω η δουλειά σας ε, για μας και στο παρελθόν ήταν πολύ χρήσιμη και οπωσδήποτε και στο μέλλον αυτό θα συμβεί. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Θα πρότεινα να περάσουμε και στο σημείο 7 και να συνδυάσουμε τη συζήτηση και για τα δύο σημεία μαζί με ρωταπαντήσεις. Κύριε Λίντσελμαν, Α έρθουμε τώρα στη μελέτη μεγατάσει στον αγροδιατροφικό τομέα, συνολική επισκόπηση και πιθανέ απαντήσεις πολιτική από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα εδώ να καλωσορίσω τη Μόνικα Πέσε και τον Ντάνιελ Τραόν. Η κυρία Πέσε είναι από ε, τον οργανισμό VVA Βρυξελών και ο κύριος Τράον από την Αρκάντια. Καθίστε στις θέσεις σας παρακαλώ. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε εξωτερικώς από την Επιτροπή Γεωργίας και νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να ακούσουμε την παρουσίαση και να δούμε τι θα συζητηθεί και στο μέλλον για, για την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Το άλλο θέμα που θα μας απασχολήσει στη συζήτηση είναι πώς στο μέλλον θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο για περισσότερους κατοίκους στον κόσμο. Πώς θα παράγουμε με τρόπο βιώσιμο τα τρόφιμα. Θα μας παρουσιάσει κάποια στοιχεία η μελέτη, τέσσερα εναλλακτικά σενάρια μεταξύ άλλων και γι' αυτό θα έλεγα Να ξεκινήσετε αμέσω κυρία Πέσκη, εφόσον το επιθυμείτε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα βάλω τα δυνατά μου για να συνοψίσω μία μελέτη 60 σελίδων μέσα σε 20 λεπτά. Ελπίζω να είναι αρκετά σαφής η παρουσίαση, ούτως ή άλλως θα ακολουθήσει η συζήτηση με υποβολή ερωτήσεων. Έτσι θα διασκεδαστούν οι απορίες σας. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Η μεγατάση στον αγροδιοτροφικό τομέα, μια γενική επισκόπηση και πιθανές απαντήσεις πολιτικής από την ευρωπαϊκή προοπτική». Η δομή της παρουσίασης. Θα κάνω ε, μια φιλομέτρηση του συνόλου της μελέτης. Θα ξεκινήσω από την εισαγωγή, δηλαδή θα εντοπίσουμε τις μεγατάσεις του αγροδιατροφικού τομέα, θα δούμε ποιες είναι οι παγκόσμιες δυνάμεις που επηρεάζουν το μέλλον της ε, διατροφικής αξιακής αλυσίδας. Θα δούμε ποια, τι γίνεται με τα τρόφιμα παγκοσμίω ε, και τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γεωργία παγκοσμίω. Θα εξετάσουμε κάποια δυνητικά σενάρια και τις συναφείς επιλογές πολιτικής ε, και θα ολοκληρώσουμε κάποια συμπεράσματα. Βάσει της ΦΑΟ και με τις παρούσες συνθήκες, μέχρι το 2050 ο αγροδιατροφικός ε, τομέας θα πρέπει να παράγει 50% περισσότερα τρόφιμα και ζωοτροφές για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ε, ανάγκες για τρόφιμα. Πολύ δύσκολος στόχος ε, να υλοποιηθεί μέχρι το 2050 και θα αυξηθεί η επισητιστική ανασφάλεια λόγω και της κλιματικής αλλαγής γιατί θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα απρόβλεπτα απροσδόκητα θα έχουμε πλημμύρες, ε, ανομβρία, τροπικές καταιγίδε, ε, κύματα καύσωνα, πυρκαγιές. Το βλέπουμε καθημερινά ήδη σήμερα. Όλα αυτά τα κρέκερικα φαινομένα θα επηρεάσουν την παραγωγή και θα επιτείνουν, θα εντείνουν τις απειλές στον κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Ας εξετάσουμε πρώτα τις μεγατάσεις που επικρατούν. Καταρχήν έχουμε εντοπίσει μία ομάδα, ένα σύνολο τέτοιων μεγάλων τάσεων. Ελπίζω να μπορείτε να διαβάσετε τη διαφάνεια, αλλιώς μπορείτε να κοιτάξετε τη μελέτη. Η σημαντικότερη μεγατάση είναι η δημογραφική τάση. Μέχρι το 2050 αναμένεται ο παγκόσμιος πληθυσμός να ανέλθει σε 10 δισεκατομμύρια. Σημαντική αύξηση λοιπόν. Ταυτόχρονα όμως θα έχουμε ε, αυξημένο κατακεφαλήν εισόδημα και αυξημένη αστιφιλία. Διαπιστώσαμε τον τελευταίο αιώνα ότι υπάρχει μια αστιφιλία μετακίνηση από την Ήπεθρο προς τις πόλεις. Επίσης, έχουμε τάσεις που αφορούν ε, το μοτίβο της κατανάλωσης. Φυσικά, η αύξηση του κατακεφαλήν εισόδηματο επηρεάζει τις ε, κατα καταναλωτικέ επιλογέ, τι του καταναλωτή. Και επίσης η αυξημένη αστιφιλία επηρεάζει τις ε, τάσεις της κατανάλωσης. Απομακρύνεται ο κόσμος από τον τόπο παραγωγής, καλλιέργειας και παραγωγής των τροφίμων και αυτό οδηγεί σε μια μεταστροφή των επιλογών του καταναλωτή και μεταστροφή στην παραγωγή. Έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή κατά κεφαλή, αυτό είναι θετικό, αλλά έχουμε και αλλαγές στο είδος των τροφίμων που καταναλώνονται και αυτές οι αλλαγές διαφέρουν ανάλογα με την ε, περιοχή του κόσμου που εξετάζουμε. Για παράδειγμα, οι αναπτυγμένες χώρες έχουν ε, φυσικά αυξημένο εισόδημα και αυξάνεται η ζήτηση ε, επεξεργασμένων τροφίμων και ε, κρέατος. Στις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες χώρες υψηλού εισοδήματο, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, έχουμε αφενός το πρόβλημα της παχυσαρκίας και υποσυτισμός λόγω της κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων σε μερικές σε μερικά τμήματα του πληθυσμού και έχουμε ακριβώς την αντίθετη τάση προς πιο υγιεινές ε, τροφές, χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη. Έχουμε φυτοφαγικά κινήματα, flexitarian, ε, ε, πανφάγων ουσιαστικά. Όλα αυτά επηρεάζουν ή τέλος πάντων φυτοφάγων που καταναλώνουν ευκαιριακά ή σπάνια σχετικά ζωικές τροφές. Όλα αυτά επηρεάζουν την παραγωγή των τροφίμων αλλά έχουμε ταυτόχρονα και άλλους, ε, άλλες αλλαγές όπως τις τη χρήση τη βιοενέργεια. Έχουμε και άλλε όμω. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Αναμένεται ότι οι, οι τεχνολογικέ εξελίξει αυξήσουν κατά 30% τις ε, σοδιές θα, θα αυξήσουν την οικολογική αποτελεσματικότητα και θα δημιουργηθούν νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Οπότε οι νέε τεχνολογικέ εξελίξει μα βοηθήσουν να υλοποιήσουμε καλύτερα το στόχο του να θρέψουμε τον κόσμο, να εξασφαλίσουμε τρόφιμα. Απ' την άλλη, έχουμε την κλιματική αλλαγή και η γεωργία ευθύνεται για μεγάλο μερίδιο των αερίων του θερμοκηπίου. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής που θα επηρεάσει αρνητικά, όπως είπα προηγουμένως, την παραγωγή λόγω των ακραίων φαινομένων ε, και θα δημιουργηθούν ίσως τεράστια προβλήματα σε ορισμένες περιοχές που ε, θα υπάρχει μεγάλη πίεση τιμών ή ε, έλλειψη προσφοράς λόγω σπα... σπάνιες τροφίμων. Επίσης, έχουμε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο φαγητού τροφίμων που χάνονται, που πετιούνται ή σπαταλώνται. Ένα τρίτο δηλαδή του της παγκόσμιας ποσότητα τροφίμων είτε πετιέται είτε σπαταλάται. Αυτή είναι τεράστια επίπτωση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απώλεια ή η σπαταλη τροφίμων. Επίσης υπάρχει ένας διαγωνισμός για, την, για τους φυσικούς πόρους. 70% του ύδατος καταναλώνεται παγκοσμίως από τη γεωργία, έχει υπολογιστεί. Κάτι που Μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσω πανίσουν οι πόροι μέχρι το 2050 και θα αυξηθεί ο, ο συναγωνισμό για την διεκδίκηση των πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή τροφίμων από τη Γεωργία μέχρι την Λιανική και φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν ε, σε ένα πλαίσιο πολιτικής και γι' αυτό ζητήσατε και τη σχετική μελέτη. Το πλαίσιο της πολιτικής το διαμορφώνουν οι διεθνείς συμφωνίες, οι πολιτικές και οι συμβάσεις που ιδεωδώς ε, συνάπτονται σε παγκόσμιο επίπεδο πολυμερές, αλλά συνήθως έχουμε και σε διμερές επίπεδο. Έχουμε την υποστήριξη της γεωργίας ε, σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στην Ευρώπη έχουμε την κοινή γεωργική πολιτική και επίσης το θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιωσιμότητας. Όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν το πλαίσιο της πολιτικής και μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τις μέγα τάσεις που σας παρουσιάσαμε. Και να δούμε τις παγκόσμιες δυνάμεις που επηρεάζουν το μέλλον της διατροφικής αλυσίδας, εντοπίσαμε τέσσερις τέτοιες παγκόσμιες δυνάμεις. Η πρώτη αφορά τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών και το πώς αυτές οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να, ε, να οθήσουν τον κλάδο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Μετά έχουμε τα οικονομικά χαρακτηριστικά της αξιακής αλυσίδας, τέταρτη δύναμη είναι η καινοτομία και στην παραγωγή τροφίμων, αλλά και στο σύνολο της αξιακής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Και έχουμε και την πραγματική μεταμόρφωση της αγοράς ε, λόγω των τεχνολογιών, των νέων τεχνολογιών. Οπότε, οι εμπορικές συμφωνίες οδηγούν σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αξιακής αλυσίδας τροφίμων στον κόσμο. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι καμία χώρα αυτάρκης ε, στην παραγωγή τροφίμων. Δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα τρόφιμα που χρειάζεται για να σητήσει τον πληθυσμό. Οπότε χρειάζεται αυτό το διακρατικό εμπόριο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου είναι ο διεθνής φορέας εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, όλες οι περισσότερες συζητήσεις γίνονται σε επίπεδο Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Αλλά πρόσφατα διαπιστώσαμε μία άνοδο των διμερών, του αριθμού των διμερών συμφωνιών που προσπαθούν να βελτιώσουν το διμερές εμπόριο μεταξύ περιοχών του κόσμου. Και είδαμε άνοδο και αυτή τη τάση. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά τη αξιακή αλυσίδα, εδώ έχουμε μία εγκάρσια ολοκλήρωση τη αξιακή αλυσίδα, τη αλυσίδα προσφορά τροφίμων, προμήθεια τροφίμων με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει αυτή η εγκαρση ολοκλήρωση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τον αυξανόμενο ρόλο των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που ίσως ενισχύσουν τις πιέσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την καινοτομία, ήδη βιώνουμε της, τον αντίκτυπο της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην παραγωγικότητα της γεωργίας και παγκοσμίω και στην Ευρώπη. Έχουμε την ε, γεωργία ακριβία, την έξυπνη γεωργία, αλλά ήδη σήμερα βλέπουμε και κάποιες καινοτομίες που δεν έχουν σχέση με την καινοτομία, αλλά με, την, ε, με τα επιχειρησιακά μοντέλα. Την ε, συνεργατική οικονομία, για παράδειγμα, και το γεγονό ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει κοινή διαχείριση κάποιων εργαλείων, κάποιων μηχανισμών στη γεωργία και έτσι στη, μπορούν να στηρίξουμε ταυτόχρονα την καινοτομία και την ε, τεχνολογική βελτίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Και έχουμε και την αλλαγή της αγοράς εργασίας. Αυτές οι ψηφιακέ πλατφόρμες παρέχουν κάποια πλούστευση τη κατάσταση και ε, βελτιώνουν την πρόσβαση των ε, πελατών στην αγορά, αλλά και βελτιώνουν και το περιβάλλον μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά ενέχουν τον κίνδυνο της μείωσης των θέσεων απασχόλησης, γιατί έχουμε αυτούς τους μεσάζοντες που διαταράσσουν κάποιο στην αξιακή αλυσίδα. Υπάρχουν λοιπόν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε αυτές τις δυνάμεις. Τώρα, να δούμε πώς αυτά τα στοιχεία προσδιορίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις για το μέλλον της γεωργίας και των αγροτικών συστημάτων, θα ήθελα να αναφέρω τρεις πυλώνες, τρεις βασικούς στόχους που επιδιώκουμε που θα έπρεπε ο κόσμος να επιδιώκει. Αφενός θέλουμε να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα της γεωργίας, αφετέρου τη διατήρηση των πόρων και την διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα της γεωργίας και θέλουμε να βελτιώσουμε τη διατροφή του κοινού και την δημόσια υγεία. Γιατί έχουμε μια αντινομία μεταξύ της, των διαφορών ασυτείας και παχυσαρκίας ε, μεταξύ των διαφορών χωρών, αλλά και της αλλαγής των διατροφικών μοντέλων. Φυσικά, η, έχουμε και άλλα φαινόμενα όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση της αστιφιλίας που πειράζουν τη γεωργία. Έχουμε την οικονομική ανάπτυξη που αυξάνει την κατακεφαλή κατανάλωση και ταυτόχρονα αυξάνει τη ζήτηση για τρόφιμα η ζήτηση αυτή θα αυξηθεί εκθετικά στο μέλλον. Κάτι που θα επηρεάσει ιδιαίτερως την ανάγκη για αύξηση και της παραγωγικότητας στη Γεωργία. Επίσης, αν οφείλουμε να αυξήσουμε την παραγωγή, η πιθανότητα κατανάλωσης μεγαλύτερων ποσοτήτων ύδατος και μεγαλύτερης χρήσης γης επίσης αυξάνεται. Έχουμε και το θέμα των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί ο αγροδιατροφικός τομέας, όπως είπαμε, ευθύνεται για αρκετές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αέριο του θερμοκηπίου. Επίσης, κατανάλωση λιπασμάτων που είναι απειλή για το περιβάλλον, αλλά και η αποψήλωση και η διάβρωση του επιφανειακού στρώματος του εδάφους είναι απειλές. Επίσης, για τη δημόσια υγεία, όπως είπα, αφενός έχουμε πείνα, σιτία και ανθρώπους ακόμη και σε ε, ε περιοχές υψηλού εισοδήματος. Έχουμε ε, ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ασυτείας λόγω της φτώχειας και ταυτόχρονα έχουμε ε, φτηνά προσιτά τρόφιμα ανθυγιεινά όμως ε, και υψηλή θερμιδικής αξίας αλλά ανθυγιεινά που ενισχύουν αυτή την αντίφαση μεταξύ παχυσαρκές και ασυτείας σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης έχουμε κάποιες χρόνιες νόσους που οφείλονται στις διατροφικές επιλογές. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη τάση ε, υγιεινής διατροφής και κύματος υγιεινής διατροφής σε κάποιες χώρες. Οπότε η διατροφή βελτιώνεται σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού, ενώ σε άλλες επιδεινώνεται. Και αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία δημιουργούν απειλές και στα θέματα της επιστημιστικής ασφάλειας. Θα εξασφαλίσουμε ε, τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε και προσιτά τρόφιμα σε ποσότητες που απαιτούνται και όπου απαιτούνται. Επίσης το θέμα της ε, ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε οι προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητα ε, που επιδιώκουμε θα ισχύουν και στο μέλλον και θα είναι προσιτά σε όλους. Και υπάρχει και το θέμα της βιωσιμότητας, της αηφορίας. Θα είναι βιώσιμη η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων και από άποψη περιβαλλοντική αλλά και από άποψη παραγωγής. Γιατί η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει και την ικανότητά μας να παράγουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και έχουμε αυτό που λέμε σήμερα την ε, ρηξικέλευθη μετατροπή της, του τρόπου παραγωγής στη Γεωργία. Αυτά που κάναμε στη μελέτη είναι να αξιολογήσουμε κάποια δυνητικά σενάρια για να προσδιορίσουμε κάποιες ε, επιλογές πολιτικής που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τα επιμέρους σενάρια. Και μάλιστα στηριχθήκαμε σε τρεις μελέτες που τις αναφέρομαι και στη, στη βιβλιογραφία που σας παρέχουμε. Έχουμε την έκθεση Lancet, το περιοδικό Lancet, ή τη, μια αντίστοιχη μελέτη για το ίδιο θέμα μιλούμε για μεγάλες εμβέλειας μελέτες που έχουν συνταχθεί για το θέμα αυτό. Κάναμε μια ανάλυση και σύγκριση αυτών των μελετών και καταλήξαμε σε τέσσερα δυνητικά σενάρια που θα τα χαρακτήριζα ως αντιφατικά. Βέβαια, ή ανταγωνιστικά μάλλον. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και άλλα σενάρια, αλλά χάρη σαφήνειας και λόγω περιορισμού των επιλογών πολιτικής που είναι πιο εύκολο να είναι αναγνωρίσιμε, εμεί εξετάσαμε τα πιο ακραία σενάρια ώστε να διαμορφώσουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το μέλλον, όπως θα διαμορφωθεί γύρω στο 2050. Οπότε θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά των τεσσάρων σενάριων. Το πρώτο είναι μικρά βήματα χωρίς στόχο όμως, δηλαδή από οικονομική άποψη ε, θα ήταν αυτό το βασικό σενάριο, το business as usual, τίποτα δεν τρέχει, καμιά αλλαγή. Οπότε κάνουμε κάποια μικρά βήματα, αλλά σε τελική ανάλυση δεν θα υλοποιήσουμε κανένα στόχο γιατί δεν έχουμε κατεύθυνση. Το δεύτερο σενάριο αφορά τη μαζική παραγωγή πάση θυσία. Δηλαδή, δίνουμε έμφαση στην παραγωγικότητα και στην παραγωγή σε αντίθεση με τη βιωσιμότητα. Αυτό που πιστεύουμε ότι είναι πιο σημαντικό είναι να ασυτίσουμε τον κόσμο και όχι να μειώσουμε την κλιματική αλλαγή. Τρίτο σενάριο είναι οι ντόπιοι επιζήσαντες. Δηλαδή, εδώ εξετάζουμε την πιθανή εξέλιξη ε, του κόσμου προς μια περιφερειοποίηση και όχι προς την παγκοσμιοποίηση. Οπότε αντί να συνεργαστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περιοχές μεμονωμένα προσπαθούν να επιβιώσουν υλοποιώντα τους τοπικούς τους στόχους. Και το τέταρτο σενάριο είναι βιωσιμότητα για όλους, που είναι το ιδεώδες και πιο ακραίο σενάριο. Ιδεώδες γιατί εδώ προσπαθούμε ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους και τη βιωσιμότητα και την ε, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αφενός και αφετέρου της παραγωγικότητας. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε τρόφιμα για όλους. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. We, um, we are from... Αρχίζουμε λοιπόν από το πρώτο σενάριο. Ορισμένες παραδοχές είναι οι ίδιες ε, σε όλα τα ε, σενάρια. Η εστίαση είναι πώς κάποιες δράσεις πολιτικής μπορούν να έχουν αντίκτυπο και να προκαλέσουν αλλαγές. Ε, δεν ε, κοιτάμε τη δημογραφική εξέλιξη, την εξέλιξη του εισοδήματος, την αύξηση και άλλα στοιχεία της οικονομίας που θα μπορούσε να επηρεάσει ε, το σενάριο. Το εξηγούμε αυτό στη μελέτη. Και όπως σας είπα, το πρώτο σενάριο είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό Ό,τι κάναμε πάντα, περιορισμένες προσπάθειες για να μειώσουμε την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Δεν αλλάζει το παραγωγικό σύστημα, το βιομηχανικό σε σχέση με το σημερινό. Καλά, έχει και λίγη καινοτομία, αλλά δεν υπάρχει ε, συγκεκριμένη και σημαντική όθηση προς τεχνολογική αλλαγή για να αυξηθεί η παραγωγικότητα οι ε, καταναλωτές ε, έχουν μια σχετική αδιαφορία ως προς το να πληρώνουν περισσότερο για ε, προϊόντα πιο υγιεινά ή φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι ανεπαρκής οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και οι πολιτικές δεν καλύπτουν θέματα ασφάλειας τροφίμων επιστηστικής. Συνεχίζουμε δηλαδή στην παλιά τακτική και πορεία. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Ποιες είναι οι επιλογές τώρα της πολιτικής, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε αυτό το σενάριο. Στην επιστηστική ασφάλεια βελτιώνουμε την παραγωγή χρησιμοποιώντας υφιστάμενα εργαλεία της ΚΑΠ στην ε, τροφική αλυσίδα χωρίς μεγάλες αλλαγές ή χωρίς έρευνα καινοτομία σε κάτι καινούριο, ότι ισχύει σήμερα. Κλιματική αλλαγή ε, αυξάνει τα κίνητρα στην πρόταση της ΚΑΠ για πιο μεγάλη αποδοτικότητα και νέες γεωργικές τεχνολογίες ε, φιλικές προς το κλίμα, αλλά και πάλι δεν είναι μεγάλες αλλαγές και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Το κάνουμε και σήμερα. Όλα αυτά είναι τύχες, Γιάννη τύχα πάντα. Ναι. Για τους αγρότες, ε, η πολιτική ασχολείται με το εισόδημά τους, το, με τις συνδεδεμένες και αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, ε, προτεραιότητες στην έρευνα και την καινοτομία ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις για την ανάπτυξη υπαίθρου, όπως γίνεται και σήμερα και οι αγρότες υποστηρίζονται από υποδομές, ας πούμε, ψηφιοποίηση, διευκολύνσεις δανεισμού, ε, εκπαίδευση νέων αγροτών ε, για να αντιμετωπιστεί το θέμα της γύρανσης του γεωργικού πληθυσμού για την ασφάλεια των τροφίμων τώρα και την ψηφιστική έχει να κάνει αυτό περισσότερο με ε, την παρακολούθηση, τον έλεγχο ότι γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε, δηλαδή εφαρμόζονται τα standards και σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές ε, χρειάζεται και εκπαίδευση ε, και για την παχυσαρκία ή τις κακές συνήθειες διατροφής και επίσης μια ευρωπαϊκή πολιτική διατροφής. Και αυτό υπάρχει ήδη. Συνεχίζουμε λοιπόν να εργαζόμαστε και να επενδύουμε στις υφιστάμενες πολιτικές. Εάν συνεχίσουμε με αυτή την τακτική, τι θα συμβεί. Η σημερινή κατάσταση θα συνεχιστεί και στο μέλλον και δυστυχώς θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα πληθυσμό που θα αυξηθεί και θα φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια στον πλανήτη και ε, η κλιματική αλλαγή θα μας αναγκάσει να αντιμετωπίσουμε ακραία καιρικά φαινόμενα αναπάντεχα που θα απειλήσουν ε, την ε, ε, ύπαρξη τροφίμων και τα αποθεματικά. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα, δεν θα μπορούμε το 2050 να θρέψουμε τον κόσμο. Και θα είναι πιο δύσκολο για μας να θρέψουμε και το σημερινό πληθυσμό, όχι πόσο μάλλον του 2050 λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επειδή αλλάζει λοιπόν ε, η κατάσταση, αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές θα επιδεινωθεί η ε, συνολική κατάσταση. Το δεύτερο σενάριο, μαζική παραγωγή πάση θυσία. Στο σενάριο αυτό ο στόχος είναι πραγματικά η μαζική παραγωγή για να μπορέσουμε να ε, θρέφουμε όσο γίνεται περισσότερο πληθυσμό. Δηλαδή όλο και περισσότερη παραγωγή για να καλύψουμε τις ανάγκες 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στη γη. Ποιος θα πληρώσει την ύφη, το περιβάλλον. Περισσότερο νερό θα χρειαστεί, περισσότερη γη, περισσότερα φυτοφάρμακα, οτιδήποτε εφόδια ε, γεωργικά για να παράγουμε και να ε, ε, παρέχουμε τρόφιμα σε 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή επεκτατική πολιτική χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τίποτα, ούτε την πολιτική, ούτε τις εταιρείες όλη η έρευνα θα είναι στο βωμό της αυξημένης παραγωγικότητας, καμία καινοτομία και τίποτα επενδύσεις για το περιβάλλον καθόλου. Επίσης, οι καταναλωτές ε, θα εστιασούν την προσοχή τους μόνο στο να τρέφονται με οτιδήποτε τρόφιμα, χωρίς να τους ενδιαφέρει το περιβάλλον. Ο στόχος λοιπόν είναι ουσιαστικά να ταΐζουμε τον κόσμο ε, σε ό,τι αφορά τις επιλογές της πολιτικής, βεβαίως στην επιστημιστική ασφάλεια, εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε ε, ε, στην ε, διαχείριση της κρίσης. Η αυξημένη γεωργική παραγωγή επηρεάζει το κλίμα και την κλιματική αλλαγή και κάνει πιο ακραία τα καιρικά φαινόμενα. Και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την παραγωγή τροφίμων. Όλα αυτά παράγουν κρίση. Ε, ξηρασία, πλημμύρες, πάγο, χιόνι, ε, ξέρω εγώ, δασικές πυρκαγιές, οτιδήποτε συμβεί θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγή και στη ζήτηση σε διάφορες περιφέρειες. Οπότε, ε, σίγουρα, για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τρόφιμα όποτε τα χρειαζόμαστε, όταν τα χρειαζόμαστε και στο επίπεδο το ποιοτικό που χρειαζόμαστε, θα πρέπει ε, να εστιάσουμε στη διαχείριση των κρίσεων. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε τις κρίσεις. Για την κλιματική αλλαγή, ο στόχος είναι να μην θεωρείται προτεραιότητα, ούτε καν να συνεχιστούν οι σημερινέ πολιτικές. Η προτεραιότητα, είπαμε, είναι η μαζική παραγωγή και αύξηση της παραγωγικότητας. Εγκαταλείπουμε τα πάντα. Ε, για τους αγρότες, ε, αύξηση της ΚΑΠ και υποστήριξη του εισοδήματός τους, γιατί στόχος πραγματικά είναι να αυξηθεί η παραγωγή. Πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή ε, και για απειρή το. Άρα και η ΚΑΠ προς αυτό το στόχο θα προσανατολιστεί και θα ε, ε, προσαρμοστεί. Θα φύγουμε από τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις και θα πάμε συνδεδεμένες, όπως το παρελθόν που διαχειριζόταν τις διατροφικές κρίσεις η Ευρώπη και αυτό φυσικά θα πρέπει να συνδέεται και με τους στόχους ε, που αναφέραμε για την επιστηστική ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός προτεραιότητας για ενημέρωση των επενδύσεων, αφού η παραγωγικότητα είναι ο στόχος και πιέζει για τη τεχνολογία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, θα πιέζουν για την έρευνα σε τεχνολογία και καινοτομία. Σε ό,τι αφορά την επισητιστική ασφάλεια, ασφάλεια τροφίμων, ε, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε ε, την τήρηση των προδιαγραφών και της ποιότητας που επιθυμούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι καταναλωτές ουσιαστικά θα εστιάσουν στο θέμα της παχυσαρκίας και του υποσυντισμού ή της κακής διατροφής και λιγότερο στη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Δηλαδή θα ενημερώνονται οι καταναλωτές για το πώς να αλλάξουν διατροφικές συνθήκες έτσι ώστε να τρέφονται καλύτερα παρά να ανησυχούν τώρα για το περιβάλλον και τέτοια πράγματα. If uh, uh, Αν δούμε λοιπόν το δεύτερο σενάριο, μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ε, να αγνοήσουμε, να παραγνωρίσουμε ή να ε, μη σπουδαιολογήσουμε όλα αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και όλες οι προσπάθειες που γίνονται για αυξημένη ε, παραγωγικότητα επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κάνουμε αυτή την προσπάθεια να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, αλλά έρχονται οι θεομηνίες και καταδικάζουν σε αποτυχία ε, αυτό το δεύτερο σενάριο, οπότε ε, επιστρέφουμε στο πρώτο σενάριο. Έρχομαι τώρα στο τρίτο. Ε, η τοπική επιβίωση, όπως την ανέφερα προηγουμένως. Ε, βασιζόμαστε στους τοπικούς παραγωγούς. Τοπικούς τώρα εννοούμε σε κάποιες περιφέρειες του κόσμου, έτσι, όχι περιφέρειες μιας χώρας. Η Ευρώπη είναι μια περιφέρεια από μόνη της. Ή ορισμένα τμήματα της Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνες τους. Γίνεται η προσπάθεια σε περιφερειακό επίπεδο. χωρίς βέβαια ακραίε εκφάνσει πούμε, να προωθούμε τα εθνικά συμφέροντα ει βάρο των περιφερειακών. Ε, λαμβάνονται περιορισμένα μέτρα για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι μια παγκόσμια προσπάθεια. Οι περιφέρειες, λοιπόν, θα θεωρήσουν ε, ότι ε, η περιφερειακή προσπάθεια είναι άσκοπη. Γιατί σου λέει, άμα εγώ κοπιάσω ιδιαίτερα και όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα, είναι μια τρύπα στο νερό. Οπότε ε, ε, ε, ε, θα πρέπει να αυξηθεί επίσης η επιφάνεια των καλλιεργούμενων Όταν κανείς προωθεί μια περιφερειακή στρατηγική, έχει στόχο την περιφερειακή αυτάρκεια ε, θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, γιατί θα είναι πιο δύσκολες και λιγότερο σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. Δηλαδή, ε, η επιφάνεια των γεωργικών γεών θα πρέπει να αυξηθεί έτσι ώστε οι περιφέρειες να παράγουν αρκετά τρόφιμα για να θρέφουν το δικό τους πληθυσμό. Βεβαίως μπορούμε να προωθήσουμε και την κοινοτομία, την αστική γεωργία και άλλες τέτοιες τάσει και μόδες ε, που ε, υποστηρίζουν και την παραγωγικότητα, αλλά για να τραφεί ο πληθυσμό θα χρειαστεί χρόνος. Ε, υγεία, τοπική παραγωγή, περιβαλλοντική προστασία, όλα αυτά είναι μια νοοτροπία και η νοοτροπία του καταναλωτή επίσης είναι στραμμένη στο τοπικό επίπεδο. Θεωρείται τον τόπιο καλύτερο και πιο υγιεινό και οι πολιτικές και εμπορικέ συμφωνίες παραμελούνται. Για την ασφάλεια τροφίμων τώρα, την επιστημιστική ασφάλεια, δυστυχώς αυτή θα αντιμετωπιστεί με ανομοιογενή τρόπο. Θα είναι μεν προτεραιότητα για την περιφέρεια με όλα τα συμπαρομαρτούντα, αλλά δεν θα είναι προτεραιότητα παγκόσμια. Και αυτό θα οδηγήσει σε δυσκολίες. Αν ξεσπάσει μια κρίση τοπική, οι άλλες περιφέρειες ε, δεν ε, θα τρέξουν να υποστηρίξουν με τις συνέπειές του. Και ε, σε ό,τι αφορά τη στήριξη και την υποστήριξη της παραγωγικότητας υπό την ε, έννοια αυτή, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι η λύση. Δηλαδή θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις και οι τεχνολογικές βελτιώσεις για να υποστηριχθεί η ε, αυτονομία και η αυτάρκεια. Η κλιματική αλλαγή, όπως σας είπα, αυτό θα σημαίνει το τέλος της παγκόσμιας προσπάθειας και θα προωθηθούν οι περιφερειακές λύσεις και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά ε, στόχος θα είναι να εξυπηρετούνται μόνο περιφερειακές ανάγκες και χώρια τοπική παραγωγή. Δηλαδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα να μην επηρεάζουν τη δική μας παραγωγή, την τόπια. Για να μπορούμε να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες της δικής μας περιφέρειας. Οι αγρότες τώρα τι θα σημαίνει για αυτούς, θα συνεχίσουν ε, την κατάσταση όπως έχει, θα διατηρηθεί η ΚΑΠ και η ενίσχυση του εισοδήματο όπως έχει σήμερα, για την ασφάλεια των τροφίμων. Ε, τα ίδια ε, με το παρελθόν, συνεχίζουμε να ελέγχουμε την τήρηση των προδιαγραφών και των προτύπων. Οι καταναλωτές βεβαίως θα προστατεύονται γιατί το σκεπτικό είναι ότι προστατεύουμε την τοπική παραγωγή, στρέφουμε τους καταναλωτές προς την κατανάλωση ντόπιων προϊόντων, αυξάνουμε τη συνειδητοποίηση του καταναλωτή, όχι όποιο και όποιο, ντόπιο. Η ασφάλεια τροφίμων και η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια ζητήματα που θέλουν παγκόσμια συζήτηση και δεν γνωρίζουν γεωγραφικά σύνορα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την κλιματική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο. Το τρίτο λοιπόν σενάριο είναι πολύ ε, απίθανο να αποδειχθεί ε, αποτελεσματικό και στα δύο επίπεδα, και στην κλιματική αλλαγή, αλλά μάλλον και στη διατροφή του πληθυσμού. Ακριβώς επειδή θα επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή η κλιματική αλλαγή και η κρίση, δεν θα φτάνουν τα τρόφιμα. Τελικό σενάριο. Το τέταρτο, τελευταίο συνεχίζουμε όλες τις δράσεις, τα συστήματα παραγωγής, ταυτόχρονα θα είναι ευφυή και αυξημένης παραγωγικότητας, αλλά και οικολογικά εστιασμένα. Δηλαδή, στόχος είναι να μειωθεί η κατανάλωση των πόρων, να μειωθεί ο αντίκτυπος μάλλον και να αυξηθεί ταυτόχρονα η παραγωγικότητα. Μεγάλη πρόκληση. Βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και των πρακτικών. Οι καταναλωτές θα έχουν μια διατροφή πιο υγιεινή και συνήθειες τέτοιες και πολιτική ενθάρρυνση όλων αυτών ε, και γίνονται επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για την υποστήριξη της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής αλλά και της παραγωγικότητας ταυτόχρονα. Με πολιτικές ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Για την ασφάλεια του τροφίμου θα πρέπει να προβλέψουμε κίνητρα στην πρόταση της ΚΑΠ για να αυξηθεί και να το η γεωργική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφιοποίηση της γεωργικής παραγωγής, ε, διάδοση της γνώσης. Η καινοτομία θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα εκεί και ως προς την παραγωγικότητα. Για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε και ε, ε, τις δεσμεύσεις μας για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και στη Γεωργία. αύξηση της ΚΑΠ για την υποστήριξη των γεωργών με ένα σύστημα αποσυνδεδεμένο και συνδεδεμένο για ειδικά προϊόντα και στόχους ασφάλειας ε, επιστηστικής θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν μια ελάχιστη επένδυση στην ε, τεχνολογία. Αυτό είναι συζητήσιμο βέβαια. Αλλά αν θέλουμε να ε, προωθήσουμε την παραγωγικότητα θα πρέπει να βρούμε νέες τεχνικές καλλιέργειας, πιο καινοτόμες. Για την ασφάλεια των τροφίμων τώρα θα πρέπει να βελτιωθούν ε, οι ποιοτικέ προδιαγραφές και να συνεχιστούν και στους καταναλωτές υποστηρίζουμε ε, την ενημέρωση και την εκπαίδευση για καλύτερη διατροφή και καλύτερες ε, διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι το σενάριο, το μοναδικό που μπορεί να μας βοηθήσει ε, να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και την πρόκληση του να έχουμε τρόφιμα για όλο τον κόσμο. Ε, επιγραμματικά, τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στη μελέτη τώρα, ε, πόσο περισσότερο θα πρέπει να παράγουμε για να μπορεί ο κόσμος να τρέφεται βιώσιμα. Έχουμε κάνει συγκριτικές μελέτες για τα σιτηρά και για το ζωικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να αυξηθεί κατά 39% η παραγωγή των σιτηρών μέχρι το 2050 ενώ ε, η κτηνοτροφία στο ζωικό κεφάλαιο λίγο λιγότερο από 30% με εστίαση στα πουλερικά. Ε, ολοκληρώνοντας λοιπόν, είδαμε ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις και προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τον πληθυσμό, με τη φύση, με τη τεχνολογία. Υπάρχουν παγκόσμιες δυνάμεις ε, και παράγοντες που είναι και ευκαιρία και πρόκληση. Ε, υπάρχουν δυνάμεις που πιέζουν προς τα πάνω και άλλες που πιέζουν προς τα κάτω. Ε, το πιθανότερο σενάριο είναι βιωσιμότητα για όλους και αηφορία με ισχυρότερα μέτρα και δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος, ε, παραγωγή ε, με βοήθεια της τεχνολογίας και πιο υγιεινός τρόπος διατροφής. Αν συμβούν όλα αυτά, δεν θα χρειαστεί το 50% αύξηση παραγωγής, όπως σας είπα στην αρχή, για να τραφεί όλος ο κόσμος. Μπορεί να αρκέσει και λιγότερο από το 50% για να ταΐσουμε το παγκόσμιο πληθυσμό. Ζητώ συγγνώμη για την ταχύτητα και μπορεί να σας ε, προκάλεσα και με μεγάλες αμφιβολίες. Είμαι έτοιμη για τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω ο συνάδελφος Ντάνιελ ε, θα έρθει εδώ ε, στο Προεδρείο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση της μελέτης. Νομίζω προκύπτουν ερωτήματα. Μπορεί κανείς να πει ότι κάποια σημεία προκαλούν ως προς την γεωργική πολιτική. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο, οπότε θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στις ερωτήσεις σας σε ένα λεπτό. Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και θα έχουμε πρώτα μετά απαντήσεις. Η κυρία Μαγκίνες πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Διάβασα την έκθεση, είμαι εδώ, κυρία μου, και να πω σε μία διαφάνεια που λέγατε να μειωθούν οι τιμές για τους καταναλωτές. Εγώ κατάλαβα ότι για να κινητοποιήσουμε την παραγωγή χρειαζόμαστε και μεγαλύτερες τιμές ε, και σε επίπεδο καταναλωτών. Αυτό θέλουμε να το συζητήσουμε και στο σενάριο 4. Μιλήσατε για την αύξηση των δαπανών στην ΚΑΠ. Όμως, θα πρέπει να δούμε σε τι βάθο χρόνου μπορεί να γίνει αυτό και για την τεχνολογία και την καινοτομία. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει για τι τεχνολογικέ λύσει, λόγω χάρη για τα γενετικώ τροποποιημένα, που κάποιε χώρε δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Θα ήθελα εδώ περισσότερε λεπτομέρειε. Και τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την παραγωγικότητα τη γεωργία και τη κοινοτροφία. Το τονίσατε και είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, όταν οργανώσαμε την ακρόαση του Αντιπροέδρου Τίμερμαν, μα είπε περισσότερη γη για τη δασοκομεία στην Ευρώπη και περισσότερο εκτατική ε, γεωργία. Ε, Κάπω μπερδεύομαι. Ω πολιτικοί θυνόντε, τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα μηνύματα τα οποία προέρχονται ακριβώ από το χώρο των πολιτικών θυνόντων. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφο Βίνο. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω όλα σε ένα λεπτό. Ξέρω ότι με μια μελέτη είναι δύσκολο να βασιστεί κανεί σε μια κλασική διαδικασία και να παρουσιάσει ταυτόχρονα και το τι πρέπει να γίνει τι κλιματικέ αλλαγέ και την προστασία μα, την ε, ε, εδαφών, ε, τη διάβρωση, την ποιότητα των εδαφών, την παραγωγικότητα, τα κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα. Όλα αυτά τα σημεία είναι όλα σημαντικά και όταν τα συζητάμε θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς πρέπει να είναι η πολιτική γεωργία. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνο δεν είναι αν θα χάσουμε κάτι από τη μία για να κερδίσουμε από την άλλη τεχνολογική κοινοτομία και, το και τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά το πρόβλημα είναι πώς αηφόρα θα μπορούμε να παράγουμε τρόφιμα και να οργανώσουμε την πολιτική γεωργίας. Δεν έχουμε βρει κάποια λύση για την αηφορία και η δική μου η πολιτική ομάδα θα ήθελε πραγματικά κάτι να κάνουμε για τον κόσμο και το περιβάλλον. Και γι' αυτό το βασικό είναι ότι θα πρέπει σε περιφερειακό επίπεδο να αξιοποιούμε καλύτερα τις διάφορες γεωργικές εκτάσεις. Στην μελέτη δεν άκουσα κάτι να λέγεται για τα οικολογικά εντατικά συστήματα όπως τα συστήματα της ε, αξιοποίησης των δασών ε, για την γεωργία. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες γεωργικής παραγωγής, αεφόρα με νόημα που μπορούν να έχουν και κοινωνική απόδοση. Ε, και για το περιβάλλον να προσφέρουν προστασία. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν κάτι περαιτέρω γι' αυτό, για το τι πρότυπα θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και να έχουμε μια αηφόρα διοργάνωση της γεωργικής παραγωγής. Γιατί αυτό είναι ο στόχος που όλοι επιδιώκουμε και, θα πρέ... και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλες τις πολιτικές ομάδες ανεξαιρέτως. Ευχαριστούμε ο συνάδελφος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παρουσίασή σας στο δεύτερο σενάριο για τη μαζική παραγωγή ε, σχέτως κόστους, μας λέτε, με κάθε τίμημα μάλλον, μας λέτε ότι αν ακολουθήσουμε αυτή την επιλογή, με τις τιμές θα που θα προκύψουν δεν θα έχουμε μαζική παραγωγή και ότι μπορεί να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις και ότι αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Με τον γάδο δεν ισχύει αυτό. Θα πρέπει να το φωνάξουμε εάν χρειαστεί Σίγουρα θα οδηγηθούμε σε ακραία ε, σενάρια εδώ. Δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερα αν δεν αλλάξουμε. Και για το σενάριο με την τοπική επιβίωση, το τρίτο, λέτε ότι κάποιες δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να ε, αναλυθούν. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ιδανικό σύστημα, αλλά σίγουρα μια περιφερειακή προσέγγιση, τοπική προσέγγιση είναι καλύτερη από αυτήν όπου παίρνουμε εκατοντάδες χιλιάδες τόνου βόηου από την περιοχή του Μερκοσούρ, εκατοντάδες χιλιάδες τόνους από την Ευρώπη τα πάμε στην Κίνα, τα στέλνουμε στη ΣΥΠΑ, παίρνουμε πορτοκάλια από την Ισπανία και τα πάμε στην Αμερική, ενώ τα πορτοκάλια της Καλιφόρνιας τα στέλνουμε στην Ευρώπη μερικές δράσεις για τον περιορισμό των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τι είναι αυτό, φαίνεται σαν ε, σενάριο όνειρο. Αφού μπορούμε να έχουμε πορτοκάλια, πατάτες και αυτά που θέλουμε σε τοπικό επίπεδο. Η ιδέα ότι δεν θα χρειαστεί μείωση λοιπόν εδώ ε, και μετά για την αύξηση της χρήσης γης. Όλοι θέλουν, μάλλον σε πολλές περιοχές, σε αυτή την περιοχή του κόσμου, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αν θέλουμε να την ονομάσουμε έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγουμε περισσότερο και από ό,τι χρειαζόμαστε. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε τοπική παραγωγή και γιατί να μην χρησιμοποιούμε λιγότερες εκτάσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ε, παράγουμε μάλλον τρόφιμα και για άλλες περιοχές του κόσμου, γιατί φροντίζουμε να μην μπορούμε να το κάνουμε μόνο τους αφού τους στέλνουμε όπλα. Ευχαριστούμε, ο κύριος Μπιτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ για αυτή τη μελέτη. Δεν θα τα σχολιάσω όλα, είπε πολλά και η Σάρα από αυτά που ήθελα να πω εγώ. Ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία που θεωρώ ουσιώδη. Την λογική που βάζει απέναντι από τη μια τη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας και την προστασία από το κλίμα. Συνάδελφε, δεν υπάρχει νομίζω μετάφραση στα γερμανικά. Κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Ε, ξαναρχίζω από εκεί που ήμουν. Ε, η λογική λοιπόν που φέρνει αντιμέτωπη την ε, δυνατότητα να παράγουμε πολύ και σε μεγάλες ποσότητες και μετά ότι όσο περισσότερο παράγουμε δεν κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή. Και υπάρχει και μια τρίτη λύση που λέει με την οικολογική γεωργία και με σωστές οικονομικές λύσεις ότι θα μπορούσαμε και να προστατευτούμε από τις κλιματικές αλλαγές και μια σχετική παθητικότητα που λέει ότι μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με 60-65% των εκτάσεων γύρω μας και να είναι παράγοντας η κατακράτηση των αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να φεύγουν στην παραγωγή. Αυτήν την λύση, αυτή την επιλογή δεν την έχετε παρουσιάσει αρκετά ανάγλυφα στη, στα σενάρια που αναπτύξατε και στην παρουσίαση της μελέτης σας. Και μετά πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε ενδεχομένω ένα άλλο μοντέλο, γιατί εμένα πιο πολύ από όλα φυσικά μου αρέσει το τέταρτο σενάριο, Περιορίζεται τις δυνατότητες επίλυσης μόνο μέσω της ΚΑΠ. Σήμερα υπάρχουν ευρωπαϊκές πιστώσεις και εθνικά κονδύλια τα οποία εκταμιεύονται και κινητοποιούνται για να αντιμετωπίσουμε τις ζημιέ που έχει επιφέρει το, το μοντέλο της άκρα της παραγωγικότητας ε, στην βιοπικιλότητα, στην εδαφική χρήση των εδαφών, ε, την ε, προστασία μας από τις κλιματικές αλλαγές, θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε κάτι περισσότερο για τη γεωργία και κτηνοτροφία και να προστατεύσουμε τους γεωργικού και τα ερχόμενα χρόνια. Δεν μπορεί μόνο η ΚΑΠ να βοηθάει προς αυτό το στόχο. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε κάπω να τηρείτε το χρονικό όριο για να προλάβουμε γέρο. Η κυρία Σάγε Πύρικ. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω εγώ μένω στην Ολλανδία και στην Ολλανδία δεν γίνεται τίποτα πια. Έχουμε τη στρατηγική για την βιοπικιλότητα, την οδηγία ε, Habitat ε, για τα, πτηνά. Δεν μιλήσατε ε, με, το, για το άζωτο καθόλου. Εμείς είμαστε ο δεύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως. Με την κατηγορία 4 έχουμε προχωρήσει. Δεν γίνεται πια τίποτα στην Ολλανδία και θα ήθελα να κάνετε μια μελέτη για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τι γίνεται με την ομοθεσία από την Ευρώπη. Αν δείτε το τέταρτο σενάριο, όλη η Ευρώπη θα έχει την ίδια νομοθεσία με την Ολλανδία. Στην πράξη όμως αυτά είναι ανεφάρμοστα. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε τίποτα πια και όλες οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να βάλουν λουκέτο. Όλα αυτά η καινοτομία που έχουμε, η έρευνα κτλ. Ε, ε, πώς θα μας βοηθήσει η Ευρώπη. Έχουν παραλύσει τα πάντα με όλη αυτή την νομοθεσία που έχουμε. Ευχαριστώ κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για τη μελέτη σας που καταδεικνύει την ανάγκη να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της επισητιστικής ασφάλειας των ε, αυξανόμενων αναγκών σε τρόφιμα και τις ανάγκης να διασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τους φυσικούς μας πόρους. Εγώ δεν έχω τόσο ερώτηση παρά σχόλιο. Βλέπουμε σε αυτό το τέταρτο σενάριο που μας αναπτύξατε ότι αυτό το τέταρτο σενάριο βρίσκεται πολύ κοντά στα ψηφίσματα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και παρά τις επικρίσεις ε, που ακούγονται, πιστεύω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε μια πραγματικά κοινή γεωργική πολιτική, ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, και θέλουμε να δώσουμε ναύσματα με οικολογικά συστήματα για καλύτερες, πιο φιλοπεριβαλλοντικές αγροτικές πρακτικές όλα αυτά που μα είπατε, εμεί τα έχουμε ήδη ψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίση δίνουμε προτεραιότητα στι επενδύσει Αφιερώνουμε 30% του δεύτερου πυλώνα στα θέματα αυτά τα φιλοπεριβαλλοντικά και επίση ε, έχουμε και άλλα μέτρα ώστε και τα προϊόντα που εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρούν τις δικές μας προδιαγραφές και τα δικά μας πρότυπα. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι εμείς ε, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω ότι και με το έργο μας θα συνεχίσουμε να είμαστε εξίσου φιλόδοξοι με το προηγούμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κατάινεν. Σας ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη αυτή. Φυσικά, ο στόχος ποιος πρέπει να είναι. Ε, να παράγουμε ε, προϊόντα υγιεινά στη σωστή ποσότητα και ε, με ακριβή τρόπο. Η τέταρτη λοιπόν εναλλακτική που μας προτείνεται είναι καλύτερη για μένα. Τι γίνεται με τους καταναλωτές όμως, θέλω να σταθώ λίγο στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Πώς μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε, να τους καθοδηγήσουμε, να έχουν τη σωστή καταναλωτική συμπεριφορά και να τρέφονται ε, με σωστό και υγιεινό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή. Ε, αυτό μας χρειάζονται οι εμπορικές συμφωνίες. Είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά. Ε, πρέπει να φτάσουμε σε μια ισορροπία. Στην Ευρώπη γίνεται έρευνα και για τα τρόφιμα. Ε, και έχει διπλασιαστεί μάλιστα η χρηματοδότηση. Έχουμε ε, καινούρια είδη φυτών, για παράδειγμα. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, αυτές οι νέες επενδύσεις να πιάσουν τόπο και να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή, όχι μόνο στην έρευνα. Και αυτό που έχει σημασία είναι το εισόδημα των γεωργών επίσης. Ε, γιατί δεν θα λάβουν υπόψη το κλίμα και το περιβάλλον οι παραγωγοί δεν μπορούν να ζήσουν. Η κυρία Αγγιλάρ. Ευχαριστώ δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την ανάγκη να αύξηση τη παραγωγή τροφίμων για έναν αυξανόμενο πληθυσμό. Βέβαια, θα πρέπει να τηρήσουμε μια οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην παραγωγή. Οπότε μπορούμε να έχουμε διαφορετικά επίπεδα, ε, μοντέλα γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να επικεντρωθούμε μόνο στο οικολογικό μοντέλο, γιατί υπάρχουν και άλλα εξίσου βιώσιμα μοντέλα για την γεωργία. Και τέτοιε μελέτες ε, μας ε, ε, συνηγορούν υπέρ του επιχειρήματος ότι θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία στη Γεωργία και να επικεντρωθούμε στις γεωργικές ε, τεχνικές και να μην μειώσουμε τους μηχανισμούς που έχουν οι Γεωργοί για να παράγουν υγιεινά και φιλοπεριβαλλοντικά τρόφιμα διαπιστώσετε ότι σε θέματα γεωργικής καινοτομίας η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σε αντίθετη κατεύθυνση από ότι οι υπόλοιπε ανεπτυγμένες χώρες. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι σημαντικό μειονέκτημα για να αντιμετωπίσουμε τις ε, παρούσες προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τη μελέτη. Έχω σημειώσει ε, τα διάφορα σενάρια, το τέταρτο βιωσιμότητα για όλους. Αυτό είναι ο παράδεισος. Ε, ωραία, τον παράδεισο καλό είναι να τον επιζητεί κανείς. Αλλά ε, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Υποθέτω ότι τίνουμε περισσότερο προς την τρίτη επιλογή. Και είπατε ότι το σενάριο αυτό έχει μειονεκτήματα, τα περιγράψατε καλά για την τόπια παραγωγή και την επιβίωση. Συμφωνείτε? Επόμενη ερώτηση. Από τη μελέτη σας, τίθεται το ερώτημα για μένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ακόμα να εξάγει γεωργικά προϊόντα ή όχι. Άλλη ερώτηση. Καινοτομία. Ωραίο ακούγεται και αυτό. Το είπε η κυρία Μαγκίνες θα ειπε η κυρια Ορίστε, μας βαίνουν και τα φώτα. Μας άλλαξαν τα φώτα από την καινοτομία. Φωτοβολταϊκά. Τι έγινε, τέλειωσαν τα φωτοβολταϊκά. τι έλεγα. Ε, καινοτομία. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε φιλικοί προς την καινοτομία. Και το τελευταίο που είπατε, ωραίο, 30% ε, της παραγωγής της γεωργικής την πετάμε, τη σπαταλάμε. Ποιο φταίει, μήπω φταίει η νομοθεσία όπου δεν φτάνει στον καταναλωτή όλη αυτή η πρωτογενή παραγωγή. Ευχαριστώ. Βλέπετε τώρα κάνουμε άσκηση για το σενάριο 4, λέει ο πρόεδρος. Ε, ε, ο συνάδελφος Ροπέ, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ. Η παρουσίαση της μελέτης ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Η μελέτη βρήθη ιδεών για το πώς ε, θα μπορούσαμε να ζήσουμε και πώς θα είναι η ζωή μετά από 30 χρόνια. Βέβαια, κατά τη δική μου γνώμη, η σημερινή γεωργία στην Ευρώπη είναι αρκετά γνωστή και παγκοσμίως και με το στάτο έχουμε πολλά προβλήματα στη Γεωργία αν δεν αλλάξουμε τίποτα. Και τα προβλήματα αυτά θα συνεχιστούν. Οπότε, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το θέμα είναι στο μέλλον τι γεωργία θέλουμε στην Ευρώπη. Βέβαια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την παρούσα κατάσταση και όλες οι ιδέες που μας παρουσιάσατε είναι ενδιαφέρουσε και μας δίνουν τροφή προσκέψη. Μιλήσατε για την ανάγκη στήριξης της γεωργίας και Είπατε επίσης ότι ίσως θα πρέπει να μεταβούμε από τις αποσυνδεδεμένες στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας αναπτύξετε αυτή σας την πρόταση. Εννοούσατε όλους τους τομείς ε, ενισχύσεων. Είμαι μόνο για τους τομείς όπου διαπιστώνουμε μια έλλειψη παραγωγής θεωρείτε ότι η μετάβαση από, τις, από συνδεδεμένες στις συνδεδεμένες ενισχύσεις θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς. Γιατί φαίνεται ότι περικόπτονται οι ενισχύσεις σε κάθε δημοσιονομική περίοδο. Και αν ε, ε, αυξήσουμε τη, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα κατά 50% χωρίς ενισχύσεις. Εσείς τι σενάρια βλέπετε για τις αγροτικές ενισχύσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Καραγιές. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Μόνικα Πέσε μας υπέβαλε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Εγώ θα σταθώ σε δύο ανησυχίε που από, τις, από το πολύ προβληματισμό που έγινε η, ε, η μελέτη. Είπατε ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, στηρίζοντα όμω την τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτομία. Επίση, είπατε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και επίσης σταδιακά να κινηθούμε προς μια βιολογική γεωργία. Δεν λέω ότι είναι τελείω ε, ασυμβίβαστη αυτή η στόχη, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα πώς θα καταφέρουμε να λύσουμε αυτή την εξίσωση που φαίνεται δύσκολη. Δηλαδή θέλουμε μια γεωργία που θα δράζεται στην βιοπικιλότητα, όπως είναι η βιολογική γεωργία, και να τη συνδυάσουμε με μια γεωργία ακριβία που θα στηρίζεται στην τεχνολογία και που μερικές φορές στηρίζεται στην ομοιομορφία. Πώς θα συμβιβάσουμε, πώς θα συμφιλιώσουμε αυτή την ανάγκη βιοπικιλότητας και μια ομοιομορφία που υπάρχει στην σημερινή γεωργία. Αυτά και σταματώ εδώ για να σεβαστώ και το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αμάρο. Ευχαριστώ. Μια παρατήρηση, χωρίς αναγκαστικά να ταχθώ υπέρ του σενάριου 4. Εδώ βλέπω κάποια σημεία συμβατότητας, είτε πω για να μην το πω έτσι, δυσκολίας. Οι μελέτες αυτές και οι συζήτησεις γίνονται για να προτιμάσουμε καλύτερα το μέλλον. Ωραία. Όμως θα πρέπει κάπου να κάνουμε μια επιλογή. Ή θα προετοιμάσουμε τη γεωργία και την κοινοτοφία του μέλλοντος στην Ευρώπη για να παράγουμε περισσότερο, ή ε, με άλλη ποιότητα και με περισσότερη ανταγωνιστικότητα, γιατί εν τέλει ε, η αγορά το επιτάσσει. Η αγορά μας είναι η ευρωπαϊκή με αγορά, αλλά και η παγκόσμια. Αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στην αγορά, διότι θα καταδικάσουμε πολλά από όσα συμβαίνουν σε επίπεδο εδαφικό, περιφερειακό και τοπικό, πράγμα που στηρίζει πολλές φορές τη γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη, σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Εάν λοιπόν η Ευρώπη πάει για μια παραγωγικότερη, ανταγωνιστικότερη, πιο καινοτόμα γεωργία και εκτενοτροφία, δεν θα, θα πρέπει να ξεχάσουμε όλους αυτούς τους τόπους όπου η γεωργία είναι πολύ, ε, πολύ πιο περιορισμένη αλλά όχι τόσο παραγωγική. Διότι θα παρατήσουμε την Ευρώπη των αγρών, αυτό όμως που εξασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη. Ναι, αλλά αυτό με το φως δεν φαίνεται να λύνεται. Έχουμε κανένα δεκάλεπτο. Φαίνεται να λύνεται, θα λυθεί μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Ε, ο κύριο Χόεσλινγκ. Καλά, μόλι πάρει το λόγο ο ε, κύριο Γιάννα, μα αλλάζουν τα φώτα και μας βαίνουν και τα φώτα. Ε, μερικά ερωτήματα δεν τα έχετε θέσει στην έκθεση. Υπάρχει μια παγκόσμια έκθεση για τη γεωργία, ε, για τη μικρή γεωργία, για την εκτατική γεωργία. Δεν μπήκατε καθόλου σε αυτό. Μιλήσατε για τεχνολογικέ λύσει. Τα τελευταία χρόνια τα ακούμε πάρα πολύ. Ο τεχνολογία θα έρθει να μα λύσει, λέει, τα προβλήματα. Το precision farming, ε, αυτό μπορεί να μειώσει το κόστος για τους αγρότες η γεωργία ακριβίας, δεν θα αυξήσει την παραγωγή. Πάνω από 20% λέτε ε, σιτηρά και περισσότερα πουλερικά. Μα το 65% των σιτηρών πηγαίνει στην ε, κτηνοτροφία. Αυτό είναι αηφορία, είναι το αντίθετο. Όλο και περισσότερο, σύμφωνα με το μοντέλο, δύο παράγουμε. Κύριε Γιάρ, στη μαζική παραγωγή βρισκόμαστε ακόμα και ε, πολύ βαθιά μέχρι τα μπούνια. Αλλά αυτό δεν είναι ούτε βιώσιμο ούτε τίποτα. Δεν αναφερθήκατε ε, ε, στα οικολογικά προϊόντα. 75% του πληθυσμού του παγκόσμιου των εντόμων έχει χαθεί. 55% των ειδών των πουλιών έχουν εξαφανιστεί. Μιλάτε για το νερό. Όχι. Μιλήσατε για την ενίσχυση της ε, έρευνας. Γιατί πάει μόνο το 1% στην οικολογική έρευνα. Μήπως αυτά τα μοντέλα πρέπει να προωθήσουμε και εκεί να κάνουμε την έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να πω ότι και τώρα που μίλησε ο κύριος Χόισλινγκ δεν ξανάναψαν τα φώτα. Ο, ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που μου έλειψε όμως είναι το πού θα μπουν εδώ οι καταναλωτές ε, γιατί το πώς θα πάει η γεωργία και η κτηνοτροφία εξαρτάται και από το τι κάνουν και οι αγοραστές και οι πολιτές. Δηλαδή, ε, αυτοί που πολλούν τα προϊόντα τους τώρα αντιμετωπίζουν πολλές πιέσεις. Μην ξεχνάμε ότι η διακύμανση των τιμών για τους γεωργούς και είναι πολύ σημαντική, ακραίων τιμών αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι με το σενάριο 2 εδώ. Συνολικά για την γεωργική μας πολιτική θα πρέπει να δούμε σε ποιο σενάριο θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Για την ασφαλή επιστημιστική παραγωγή και για ολόκληρο τον πληθυσμό του κόσμου θα πρέπει ποιες, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα προταθούν και θα επιλέξουμε. Äh, Ευχαριστούμε. Κρίστανσον. Σα ευχαριστώ. Σίγουρα. Είναι κρίμα που έχουμε τόσο σημαντική απώλεια και σπατάλη τροφίμων, 30% το 1 τρίτο σχεδόν. Ε, αυτό είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις που καλούμαστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Επίσης έχουμε αύξηση του πληθυσμού μέχρι το 2050. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ελπίζουμε οι νέες τεχνολογίες να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή αλλά και την ανάγκη πιο βιώσιμης παραγωγής. Αλλά αν αυξήσουμε την παραγωγικότητα θα πρέπει να το κάνουμε χάρη στις ε, νέες τεχνολογίες και αυτές να εκμεταλλευτούμε. Σίγουρα οι νέες τεχνολογίες θα μας βοηθήσουν και να αυξήσουμε την, παραγωγικο, παραγωγικότητά μας αλλά και να τηρήσουμε μια βιωσιμότητα. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα σενάρια, νομίζω ότι θα μπορούσαμε ε, ακόμη και να τα συνδυάσουμε και φυσικά κάθε ήπειρος είναι διαφορετική. Μιλήσατε για τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην κοινή ακροτική πολιτική, αλλά και στην ε, διατροφική αλυσίδα. Σε αντίθεση με εσά, εγώ πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση δεν θα περάσει μόνο από τα μαζικά, από τα μαζικά δεδομένα, αλλά θα χρησιμοποιηθεί και στην γεωργική παραγωγή. Οι τεχνολογίες ε, και τις επικοινωνίες και τις πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στη γεωργία και κυρίως να κρατήσουμε ζωντανή την Ήπεθρο, να μην απεριμωθεί. Γιατί στην Ήπεθρο έχουμε γεωργία και κτηνοτροφία, εκεί παράγονται τα τρόφιμα. Μα είπατε ότι το 70% του πληθυσμού στο μέλλον θα ζει στι πόλει. Οπότε πότε, πώς θα εξασφαλίσουμε ψηφιοποίηση και τη υπαίθρου, πώς θα φτάσει το ευρυζωνικό διαδίκτυο και στι αγροτικές περιοχέ. Αν δεν έχουμε ψηφιοποιήσει και στην Ήπεθρο, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απερίμωση και εγκατάλειψη και αστιφιλία. Οπότε σίγουρα θα μειωθεί η γεωργική παραγωγή. Η προστασία των μικρών εκμεταλλεύσεων είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε το ίντερνετ, το διαδίκτυο, η ψηφιοποίηση να φτάσει στην Ήπεθρο για να μπορεί ο κόσμο να διαβεί εκεί. Ευχαριστώ. Ο κύριο Δεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, προσκεκλημένους μας για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Οπωσδήποτε, μια και μιλάμε για κλιματικές αλλαγές, η γεωργία και η είναι μέρος του προβλήματος. Ίσως δεν το τονίσαμε αρκετά ότι θα μπορούσε να είναι ε, και μέρος της λύσης και είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό. Ε, σκεφτείτε τι θα γίνει με περιβαλλοντικές πολιτικές, πολιτικέ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που να μην περιλαμβάνουν γεωργού και κτηνοτρόφου. Είναι αδιανόητο. Εδώ λοιπόν να σκεφτούμε τις προοπτικές επανεθνικοποίησης της μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η πρόταση που συζητάμε μάλλον είναι αν θα επιλέξουμε μεταξύ τρίτου και τετάρτου σεναρίου. Και εδώ θέλω να προκαλέσω λίγο με την ερώτησή μου. Νομίζω πιο σωστό είναι να πάμε προς το τρίτο ε, σενάριο, ε, να αφήσουμε περισσότερη ελευθερία στα κράτη-μέλη και όχι προς το τέταρτο, αυτό που από ό,τι ακούσατε υποστηρίζουμε εμείς περισσότερο. Νομίζω ότι πάμε σε σωστή κατεύθυνση, γι' αυτό και για το φως. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μπούντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω τη μελέτη αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μας επιτρέψει μέσω μακροπρόθεσμα να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Έχω μια ερώτηση για τις σπατάλη τροφίμων. Πουθενά σε κανένα από τα τέσσερα σενάρια να αναφέρεται έχουμε περιορισμούς και μεγάλους ε, ως προς τους πόρους για την παραγωγή. Ένας ε, στόχος πάρα πολύ σημαντικός είναι να μειώσουμε τις πατάλη τροφίμων. Φυσικά δεν φτάνει μόνο αυτό. Ε, θα πρέπει να έχουμε μικρές αλυσίδες τροφοδοσίας έτσι ώστε να προλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο της πατάλης και να παρέχουμε και τρόφιμα ε, που έχουν παρεχθεί με μικρή παραγωγή χαμηλή διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές οι βραχίες αλυσίδε ταυτόχρονα μας επιτρέπουν να προστατεύουμε το περιβάλλον. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Κάστρο που ε, μίλησε για τους αγρότες ότι θα πρέπει να αμείβονται για την προστασία του περιβάλλοντος που παρέχουν. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η παχυσαρκία και θα πρέπει να εντείνουμε τις πολιτικές πρόληψης ε, της παχυσαρκίας. Ταυτόχρονα όμως να ενθαρρύνουμε την ε, κατανάλωση ε, βιολογικών προϊόντων, βιολογικών τροφίμων, που είναι και υγιεινά για τον καταναλωτή, αλλά και ε, επιτρέπουν να καταναλώνει λιγότερα φάρμακα. Το έχετε σκεφτεί αυτό το θέμα της παλάτης. Ε, σπατάλης, ε, Γκερέρο. Ευχαριστώ. Τρία σχόλια σύντομα. Καταρχήν, μία ανησυχία. Πώς αναλύονται τα στοιχεία, γιατί νομίζω ότι δεν είναι πολύ μεροληπτική η μελέτη προς τα σενάρια που επιλέγει. Δεύτερον, έχουμε από το είπες και από, το IPCC παρόμοια σενάρια με, τις με την κλιματική αλλαγή να δημιουργεί πολύ πιο ακραία σενάρια. Αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη η σχετική μελέτη, η δική σας μελέτη. Υπάρχουν στοιχεία που μας αποδεικνύουν ότι οδεύουμε προς ένα κλιματικό χάος. Δεν φαίνεται να λαμβάνετε τόσο σοβαρή κατάσταση υπόψη στη μελέτη σας. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα την περιορισμό της πατάλης τροφίμων, γιατί 30% των ε, τροφίμων πετιόνται. Ενώ μιλήσετε για περισσότερη παραγωγικότητα, ένα εκτάριο, περισσότερη κατανάλωση, αλλά ε, δεν ε, επικεντρωνόμαστε στο απολύτως απαραίτητο που είναι να διορθώσουμε αυτή τη σπατάλη τροφίμων, που είναι το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων. Επίσης, έχουμε ε, τεράστια κατανάλωση φυσικών πόρων από την κτηνοτροφία. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη για να κάνουμε μια πιο μεγάλη εξοικονόμηση των πόρων. Και φυσικά να αλλάξουμε τα καταναλωτικά μας μοντέλα που μερικές φορές ε, συμβάλλουν σε αυτή την κατασπατάληση των τροφίμων. Ευχαριστώ. Κύριε Τολαρίν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σας που διάβασα με μεγάλη χαρά. Σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές προκλήσεις και την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ε, θα ήθελα κάποια επιπλέον στοιχεία. Ε, οι νέοι κάτοικοι του πλανήτη κάπου θα πρέπει να διαβιώνουν. Τι προβλέπετε στα διάφορα σενάρια για να μην χάσουμε ε, μεγάλες επιφάνειες που έχουν και γεωργικό δυναμικό, αλλά και θα, ταυτόχρονα θα πρέπει να στεγάσουμε τον νέο πληθυσμό. Το 2050 δεν είναι και τόσο μακριά. Αν συνεχίσουμε την ΚΑΠ, ε, θα έχουμε όλο και περισσότερες διαμαρτυρίες κατά των γεωργών. Μερικέ φορές οι καταναλωτέ μετατρέπονται σε καταγγέλλοντε, σε δημοσιογράφους ή έτσι νομίζουν τουλάχιστον και φαίνεται ότι η αστιφιλία τους απομάκρυνε από την Ήπεθρο και του απομάκρυνε και από το γεωργικό επάγγελμα που δεν το καταλαβαίνουν. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε σε μια τράπεζα να συγκαλέσουμε και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους γεωργούς, εκπροσώπους των καταναλωτών, ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους μέχρι το 2050 και να γίνουν αντιληπτές συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για τη γεωργία και να τις συζητήσουμε όλοι μαζί από κοινού. Επίσης, ό,τι αφορά την καινοτομία, μέχρι πού είμαστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να πάμε. Για παράδειγμα, όλοι συμφωνούμε ε, για την καινοτομία σε ό,τι αφορά ε, την βιολογική γεωργία που χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα φυτά για να περιορίσουμε την ε, κατανάλωση φυτοφαρμάκων γιατί λειτουργούν ως ζυζανιοκτώνα ή απορροφούν κάποια παράσιτα. Μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι λοιπόν να πάμε στην καινοτομία. Ο κύριος Ρούσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη σαφέστατη παρουσίαση σε ό,τι αφορά τη σπατάλη τροφίμων, food waste λέγεται αυτό στα αγγλικά, είπατε στην παρουσίασή σας ότι το 1 τρίτο της παραγωγής τροφίμων ε, σπαταλάται υπετιέται; Ποια, ποιος είναι ο ορισμός του waste εδώ της σπατάλης. Το 1 τρίτο μου φαίνεται τεράστιο ποσοστό. Ε, ε, αν κοιτάξουμε τη γεωργική παραγωγή, υπάρχουν πάντα παραπροϊόντα, υποπροϊόντα, τα οποία εκμεταλλευόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Εάν μπαίνουν όλα αυτά στην κατηγορία σπατάλη τροφίμων, φυσικά αυξάνεται το ποσοστό. Μπορείτε παρακαλώ να ορίσετε τη σπατάλη τροφίμων, πόσο ευρύ είναι αυτός ο ορισμός. Και δεύτερη ερώτηση, σε ποιο κρίκο της αλυσίδας χάνονται τα περισσότερα τρόφιμα, ποιος πετάει, ποιος παταλάει, ο καταναλωτής ή ο Γεωργός ή στην ε, ε, αλυσίδα παραγωγής μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα. Το ξέρω ότι είναι πολύ ειδική ερώτηση, αλλά θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες στην απάντησή σας. Ευχαριστώ. Ε, ο συνάδελφος Ντεσέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ντεσέρλα. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ο κύριος Χόισλινγκ προηγουμένως μίλησε για την εξαφάνιση ορισμένων εντόμων και της βιοπικιλότητας ε, κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει ένα άλλο είδος υποεξαφάνιση που δεν ε, αναφέρουμε πολύ συχνά που είναι οι αγρότες και οι αγρότησες. Στην Ευρώπη έχουμε φιλοδοξίες για τα γεωργικά αλλά είμαστε οι μόνοι που χάνουμε τόσο πολλούς αγρότες και αγρότησες. Είναι καταστροφική η δημογραφική εξέλιξη και θέλω να σας ρωτήσω πέρα από τα τέσσερα σενάρια που μας παρουσιάσατε μήπως θα μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιου στόχους. Είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους χάνοντας τόσους αγρότε και αγρότησε. Και μια απάντηση για να φτάσουμε στους στόχους μας και ε, στις φιλοδοξίες για το περιβάλλον, η λύση είναι το εισόδημα, υπόθηκε αυτό, εισόδημα γεωργικό στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δυστυχώς σήμερα οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν αρκεί, δεν φτάνει σε αυτό το στόχο. Ε, για να έχουμε σταθερότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται εκβάθρον λύσεις στη μελλοντική ΚΑΠ που θα πρέπει να προτείνουμε εμείς αύριο. Ευχαριστώ, συνάδελφος Λεμπρετόν. Ευχαριστώ για τη μελέτη. Τέσσερις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη αναφερθήκατε στο ορίζοντα του 2050 αύξηση του παγκοσμίου εισοδήματος κατά κεφαλή. Αυτό πραγματικά με εκπλήσει πάρα πολύ γιατί είναι τελείως ετερογενεί οι καταστάσεις. Ποια είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία που σας επιτρέπουν να ισχυρίζεστε κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση. Είστε υπέρ του σεναρίου 4. Αυτό είναι ο, ο ύμνος στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και στην απελευθέρωση των, των αγορών. Σωστά το κατάλαβα. Τρίτον, ε, ε, είναι μια καρικατούρα το σενάριο 3 και το ειρωνεύεστε και από τον τίτλο, αλλά δεν αναφέρεστε στις αρετές, ε, ε, οι βραχίες αλυσίδες που είναι βιώσιμοι. Επίσης, ο σεβασμός ε, της επιστημιστικής κυριαρχίας που ζητάει ο κόσμος. Από την άλλη, αντίθετα λέτε ότι δεν θα υπέρχουν διεθνή φόρα για την κλιματική αλλαγή. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο συστηματικά φέρνετε αντιμέτωπο το τοπικό στοιχείο και την τοπική παραγωγή με τη βιωσιμότητα. Τέταρτον, πολύ λίγο αναφερθήκατε στους αγρότες. Τι γίνεται με την οικογενειακή γεωργία στο σενάριο που ονειρεύεστε το υπαριθμό 4. Ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αποφασιστική ερώτηση. Πόσο γίνεται με λιγότερου πόρου, με τρόπο αηφόρο να θρέψουμε περισσότερο κόσμο στον πλανήτη. Και βεβαίω αυτό που προκύπτει είναι κάτι το πραγματικά αξιοσημείωτο πώς θα πρέπει να αποδεχτούμε και την αλλαγή στη σοδιά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε, στο ρόλο, στο μέλλον, τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι πολυεθνικές αυτές που θα διαχειρίζονται τη γεωργική παραγωγή. Είναι σημαντικό και δεν έχει απαντηθεί. Και τρίτον, τι γίνεται με τη χρήση της γης σε σχέση με τη γεωργική παραγωγή, για την παραγωγή τροφίμων, την ε, ε, διακομιδή των αποβλήτων και το τι γίνεται με τα απόβλητα που παράγονται και τη σπατάλη των τροφίμων. Βλέπουμε ότι το 40% τη σπατάλη οφείλεται στα... Ε, γιατί το 40% τη σπατάλη ευθύνονται τέτοια τα νοικοκυριά στη Γερμανία, παραδείγματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα διακινήσουμε αυτό με τρόπο αηφόρο. Uh, Ευχαριστώ και λυπάμαι για την πληθώρα των ερωτήσεων. Μία μελέτη κάνατε, δεν είστε αρμόδιοι να απαντήσετε σε όλα αυτά. Δεν είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι το τέταρτο σενάριο είναι ο παράδεισος, αλλά ότι τα τρία προηγούμενα είναι η κόλαση. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πέμπτο σενάριο που να είναι πιο εφικτό. Γιατί μιλήσατε για την ρηξικέλευθη ε, μεταστροφή σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Αυτό από πού προέκυψε, από τη μελέτη Lancet Επίσης, πολλά λέτε για τα τρόφιμα, για τους γεωργούς. Για την ελιά όμως δεν λέτε τίποτα, για, το, για τα ψάρια. Γιατί και η πρωτεΐνη που λαμβάνουμε από τους ωκεανούς ε, εντάσσεται στο σύστημα. Δεν αναφερθήκατε όμως καθόλου σε αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ. Ε, τελευταίος ο συνάδελφος Ντάβιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα είναι αν έχουμε ακολουθήσει και ως τώρα τη σωστή κατεύθυνση. Ε, πρέπει να δώσω το εξή παράδειγμα ε, για τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ε, πριν από 30 χρόνια ήμασταν αυτάρκης ε, ως προς την παραγωγή των τροφίμων. Τώρα είμαστε αυτάρκης ως προς 38%. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε πόσο έχει μειωθεί κατά ένα τέταρτο η παραγωγή μας είναι καλό αυτό, είναι κάτι το θετικό. Την παραγωγή τη χειρίζεται οι πολυεθνική όμιλη πιέζουν τις τιμές και πέφτει η ποιότητα. Είναι κάτι το σωστό αυτό, είναι αυτό που θέλουμε. Έχουμε τέσσερις φορές λιγότερες επιδοτήσεις από το Βέλιο και τις κατοχώρες και πρέπει να ζήσουμε με την κοινή αγροτική πολιτική και συνεχίζω να ακούω ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Μήπως κάπου πρέπει να κάνουμε και λίγο πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε με τον κύριο των ερωτήσεων. Θα ήθελα το λόγο ίσως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Χανιώτης, δεν ξέρω αν το είπα σωστά. Αν γίνεται λίγο σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να, με, να σχολιάσω σε αυτή τη συζήτηση. Η σύνοδος για τους ε, νέους γεωργούς θα επικεντρωθεί στην ε, γεωργία από την παραγωγή στην κατανάλωση, από το χωράφι στο πιάτο του καταναλωτή. Τα τέσσερα σενάρια τώρα αυτά που είδαμε είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Εγώ να επικεντρωθώ σε αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει ήδη. Πρώτα απ' όλα, όλο και περισσότερο φαίνεται ότι το τομέα παραγωγής τροφίμων ε, βασίζεται στη ζήτηση. Και βεβαίω είναι πολύ ετερογενεί οι παράγοντε που επηρεάζουν τη ζήτηση. Αλλάζουν οι προτιμήσει και τα γούστα των καταναλωτών. Και πολλέ φορέ στον ανεπτυγμένο κόσμο αυτό βγαίνει και στα πρωτοσέλιδα. Και βεβαίω το επίπεδο παραγωγή που απαιτείται από του κτηνοτρόφου και γεωργού αλλάζει. Λιγότερο κρέα και πώ επηρεάζεται και πώ παράγεται, μάλλον ενδιαφέρει περισσότερο. Αλλά μεγάλα μέρη ε, του πληθυσμού του κόσμου δίνουν σημασία στι τιμέ. Έχει σημασία το πόσο ακριβά είναι τα προϊόντα προϊόντα. Και αυτό επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο και τους, τα μοτίβα κατανάλωσης. Ε, δηλαδή, το πώς ε, αλλάζουν ε, οι σχέσεις με τα προϊόντα. Στον ανεπτυγμένο κόσμο τα τελευταία 15 με 20 χρόνια λόγω χάρη το βόλιο κρέας καταναλώνει το όλο και λιγότερο. Στον αναπτυσσόμενο όλο και περισσότερο. Και έχουμε διαφορές και σε άλλους τέτοιους τομείς. Αναφέρθηκα στο βόλιο γιατί είναι αυτό που βγαίνει στα πρωτοσέλιδα. Επίσης, ε, άλλες σημαντικές αλλαγές υπάρχουν στη διατροφική αλυσίδα. Λόγω χάρη αυτό που έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες των λιανοπολιτών για τα βιώσιμα τρόφιμα. Όλα αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν το αν χρειαζόμαστε περισσότερα και η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Ναι, θα χρειαστούμε περισσότερα, ακόμη και για τον απλό λόγο ότι ο πληθυσμό του κόσμου θα αυξηθεί ε, στο μέλλον από σε σχέση με το σήμερα. Και βεβαίω θα δούμε τι εισόδημα κατά κεφαλήν μπορεί να υπάρξει. Και τώρα για του σχετικού παράγοντε που επηρεάζουν, διότι υπάρχουν δύο αντικρώμενε δυνάμει εδώ που δρούν. Πρώτα απ' όλα αυτέ που επηρεάζουν το κόστο παραγωγή. Οι κλιματικέ αλλαγέ είναι ο πρώτο παράγοντα, διότι προκαλεί σοβαρότατε δυσκολίε σε πολλά μέρη του κόσμου ε, με τις αλλαγές τους κλασικούς τρόπους παραγωγής που είχαν συνηθίσει ω τώρα γεωργικοί κτηνοτρόφοι. Και δεύτερον, το, η αύξηση του κόστους παραγωγής, ιδίω στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, τα πρότυπα μάλλον, για την ε, ε, μη σπατάλη των τροφίμων, τα περιβαλλοντικά, τα οικολογικά. Και μετά υπάρχουν σαφές, σαφείς πιέσεις από τη χρήση της ενέργειας στη γεωργία, ε, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη χρήση της γης ή το πώς ε, επηρεάζουν οι ζωοτροφές. Έχει και αυτό να κάνει με το κόστος. Ταυτόχρονα, Υπάρχουν πολύ σημαντικοί παράγοντες που βοηθούν να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Θα μπορούσαμε να τους συνοψίσουμε στον όρο γεωργία και κτηνοτροφία 4,0, 4.0 να πω σύντομα ότι ως τώρα η αναλογία ζήτησης και προσφοράς δεν είναι κάτι που παρατηρούμε μόνο σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά παγκοσμίω και προκαλεί αβεβαιότητας και ανασφάλεια, όχι μόνο λόγω της διακύμανσης στις τιμές, ε, κάτι στο οποίο είναι συνηθισμένη η γεωργική αλλά και το επίπεδο των τιμών. Σε τι τιμές θα πουλάνε μακροπρόθεσμα οι γεωργικοί κοινοτρόφοι. Και Τρίτο και τελευταίο σημείο εδώ για την Γεωργία 4,0, τη νέα γενιά της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Είναι αλήθεια ότι η προηγούμενη μεγάλη μεταμόρφωση του αγροδιατροφικού τομέα ονομάστηκε Πράσινη Επανάσταση. Όμως το αποτέλεσμα είναι πολύ σαφές. Μας επιτρέπει να, να αντιμετωπίσουμε οικονομικά προβλήματα αυξάνοντας την παραγωγικότητα, κοινωνικά αυξάνοντας την παραγωγή τροφίμων και έχει και μια σχετική προστασία του περιβάλλοντος μέσα. Ε, χρειάστηκε μια γενιά για να το καταλάβουμε, αλλά το νιώθουμε ήδη. Τώρα με τη γεωργία της νέα γενιάς τι καταλαβαίνουμε ότι δίνει την δυνατότητα να αυξήσουμε ταυτόχρονα και την οικονομική αποτελεσματικότητα με μεγαλύτερη παραγωγικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος να την κάνουμε αποτελεσματικότερη με πολύ μεγαλύτερη, μικρότερη μάλλον ένταση στις προσπάθειες. Όμως ασκεί μεγάλες πιέσεις στην κοινωνική συνιστόσα. Τα δημογραφικά, το κενό μεταφορά τα κενά και τα χάσματα στη μεταφορά γνώσεων διαγενειακά. Όμω μπορεί να δημιουργούνται και περισσότερε ευκαιρίε, διότι αυτέ οι τεχνολογίε είναι ουδέτερε ω προ τον αντίκτυπο που, που επιφέρουν, ε, αλλά όχι ω προ τη συνεργασία μεταξύ γεωργών ή τη μεταφορά γνώση που απαιτείται. Το τι θα κάνουμε λοιπόν θα εξαρτηθεί από το τι αριθμού ε, θα χρησιμοποιήσουμε ω θεμέλιο για τι αποφάσει μα, για τι έκπομπε των αερίων του θερμοκηπίου, για τι πατάλη των τροφίμων και ούτω καθεξή. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του τι πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί για το ποια είναι η βασική γραμμή, η γραμμή αφετηρία από την οποία θα ξεκινήσουμε και εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε ευκαιρίες και στο μέλλον να συζητήσουμε από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πέσκε, θα πρέπει να βρείτε την υψηλή τέχνη της ε, συμπερίληπτης απάντησης σε 25 από αυτές τις ερωτήσεις στο σύντομο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Τα 11 λεπτά που μένουν. Έχετε το λόγο. Ανέφικτη αποστολή. Εν πάση Mission impossible. Το πρώτο σχόλιο που σημειώσα είναι ότι το γεγονός ότι λαμβάνουμε τόσα σχόλια και τέτοια πληθώρα ερωτήσεων, καταιγισμός πραγματικός, δείχνει ότι η μελέτη που όπως σας είπα στηρίζεται σε σενάρια που είναι ακραία. Εμείς τα επιλέξαμε έτσι και αντικρουόμενα και ανταγωνιστικά. Και ακριβώς αυτό δημιούργησε την ζωήρη συζήτηση. Εμείς προτείνουμε κάποια σενάρια φυσικά, αλλά το σημείο φετηρίας είναι ότι η επιλογή των σενάριων εσκεμμένα ήταν αυτή για να είναι ακραία τα σενάρια και πολύ ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Σίγουρα υπάρχουν και πιο ενδιάμεσα σενάρια, αλλά επίτηδε διαλέξαμε τόσο ακραία σενάρια για να εστιάσουμε την προσοχή σας σε πιο ακραίες περιπτώσεις. Και τελικά φαίνεται ότι το καταφέραμε. Μερικά από τα σχόλια και οι απορίες σας ε, σχετίζονται περισσότερο με πολιτικές αποφάσεις ή αποφάσεις πολιτικής. Και αυτές τις ε, ερωτήσεις δεν μπορώ να τις απαντήσω εγώ, γιατί εμείς είμαστε ανεξάρτητοι σύμβουλοι. Προσπάθησα να ομοδοποιήσω κάποιες ερωτήσεις και σχόλια, κράτησα σημειώσεις και ελπίζω να καλύψω τις περισσότερες. Ένα σχόλιο, μια ομάδα σχολείων αφορά τη σπατάλη των τροφίμων. Μας προσάψατε σχετική αδιαφορία, ότι δεν το αναλύσαμε δεόντως. Αλλά είχαμε μόνο 20 λεπτά, δηλαδή 10-12 διαφάνειες. Λογικό ήταν να μην έχουμε διεξοδικό κείμενο. Η κυκλική οικονομία αναφέρεται στο σενάριο, στο τέταρτο σενάριο, αλλά όχι μόνο στο τέταρτο σενάριο. Συμφωνώ απόλυτα ότι η σπατάλη των τροφίμων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το 1 τρίτο των τροφίμων πετιέται, το σπαταλάμε. Είναι τεράστιο αυτό το ποσό. Τεράστια ποσότητα και σίγουρα η βελτίωση της σπατάλης των τροφίμων θα βελτιώσει τη γενικότερη κατάσταση. Και θα πρέπει να δούμε πού εντοπίζεται αυτή η σπατάλη τροφίμων. Νομίζω ότι σε όλες σε όλους τους κρίκους της αξιακής αλυσίδας υπάρχει σπατάλη τροφίμων. Γιατί η απώλεια τροφίμων, η σπατάλη τροφίμων δεν εξετάζεται μόνο ε, στην αποχώρηση των προϊόντων από το χωράφι μέχρι όσο φτά, μέχρι φτάσουν στη μεταποίηση. Υπάρχει φθορά τροφίμων ακόμη και στη μεταφορά των τροφίμων. Επίσης, έχουμε αγορά τροφίμων στα σούπερ μάρκετ και πολύ συχνά, το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, έχουμε υπέρβαση ημερομηνία λήξης τα τρόφιμα που έχουν περάσει την ημερομηνία λήξη πετιώνται. Αυτό είναι κακικός προγραμματισμός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ίσως. Ή μερικές φορές έχουμε σπατάλη τροφίμων γιατί μερικές φορές εσκεμμένα καταστρέφονται τρόφιμα για να μείνουν σταθερέ οι τιμέ του. Επειδή η μεγάλη προσφορά τροφίμων στην αγορά οδηγεί σε μείωση των τιμών. Γι' αυτό μερικέ φορέ καταστρέφουμε τρόφιμα για να διατηρήσουμε υψηλά τι τιμέ. Οπότε για πολλού και διάφορου λόγου έχουμε πέταγμα σπατάλη τροφίμων. Και σίγουρα το θέμα αυτό θα μπορούσαμε να το πραγματευτούμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση και είναι από τα βασικά στοιχεία της έκθεσης. Μπορεί να μην αναφέρθηκε αρκετά στις διαφάνειες, αλλά και οι διαφάνειες αναγκαστικά ήταν μια σύνοψη της μελέτης. Πριν περάσουμε σε άλλο θέμα, θα ήθελα ο συνάδελφος να σας μιλήσει για την καινοτομία. Ναι. Ευχαριστώ, Μόνικα. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν την καινοτομία και το είδος της καινοτομίας που θα πρέπει να αναπτύξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, την τελευταία δεκαετία έγιναν τεράστιες προσπάθειες ώστε ξεπεράσουμε τη συμβατική γεωργία και να περάσουμε σε άλλα είδη γεωργίας όπως τη βιολογική. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι αυτές οι αλλαγές ε, αναμένονται από όλους τους ε, παράγοντες της αξιακής αλυσίδας ε, από τους παραγωγούς μέχρι τους καταναλωτές. Ναι, όντως όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας θέλουν την καινοτομία αλλά η πρόοδος είναι αρκετά αργή. Αυτή είναι μια παρατήρηση και έχουμε εδώ ένα βασικό στοιχείο της καινοτομία. Η καινοτομία δεν θα πρέπει να είναι μόνο τεχνολογική, αλλά και κοινωνική. Δηλαδή, αυτό που παρατηρήσαμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια είναι ότι σήμερα οι καταναλωτές είναι πιο θετικοί απέναντι στην καινοτομία, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Στο παρελθόν οι ερευνητές ε, ε, πρότειναν καινοτόμε τεχνολογίε τι χρησιμοποιούσαν ίσω οι γεωργοί, αλλά οι καταναλωτέ δεν είχαν λόγο στη διαδικασία αυτή και στην ε, αποδοχή της καινοτομία. Κάτι που δεν ισχύει πια. Οι καταναλωτές πια συμμετέχουν στη συζήτηση για τις γενετικώς τροποποιημένες τροφές, για τα φυτοφάρμακα, για τα χημικά προϊόντα. Είναι πιο ενεργοί και πιο δραστήριοι και συμμετέχουν περισσότεροι καταναλωτές. Οπότε θέλουμε ε, όταν οι καινοτομίε γίνονται αποδεκτέ, να γίνονται δεκτέ από όλου του κρίκου τη αξιακή αλυσίδα και από του καταναλωτέ. Και αυτό σήμερα ισχύει. Γίνονται πιο αποδεκτέ οι καινοτομίε, γιατί οι καταναλωτέ είναι πιο ενεργοί και ενημερώνονται πολύ καλύτερα για το λόγο δημιουργίας της καινοτομία και εφαρμογής της καινοτομία. Οπότε μπορούν να την ασπαστούν πιο εύκολα οι καταναλωτές γιατί είναι καλύτερα κατατοπισμένοι. Θα πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνει πραγματικά ο καταναλωτής όλες τις επιμέρους πτυχές του θέματος. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα μηνύματα να είναι σαφή και να μεταδίδονται με σωστό τρόπο στον καταναλωτή, ώστε ο καταναλωτής που θα κάνει και την τελική επιλογή να έχει ξεκάθαρα μηνύματα και καλή ενημέρωση για να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Και αυτό θα είναι βασικό στοιχείο για την αποδοχή της καινοτομίας. Θα πρέπει να γίνεται σωστή διάδοση των πληροφοριών για την καινοτομία. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές τώρα σχέσεις, πολύ σημαντική είναι η θέση του γεωργού στην αλυσίδα τροφοδοσίας. Γιατί φάνηκε από τις συζητήσεις με τους καταναλωτές ότι οι καταναλωτές ε, δεν λαμβάνουν καν υπόψη τη θέση του γεωργού στην αλυσίδα ε, ανεφοδιασμού. Θα πρέπει να επαναφέρουμε, να αποκαταστήσουμε τη σωστή θέση του Γεωργού στην αλυσίδα ανεφοδιασμού. Μάλιστα. Κάποιες σύντομες απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Ποια ήταν ε, η πηγή που χρησιμοποιήσαμε για την αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματο. Το ΦΑΟΣΤΑΤ. η στατιστική υπηρεσία της ΦΑΟ και στη μελέτη έχουμε σχετικές λεπτομέρειες. Η περιοχές υψηλού εισοδήματο θα μειωθούν στο μέλλον ε, του κατακεφαλήν εισοδήματο. Γιατί στις ανεπτυγμένες χώρες αυξάνονται αυτές οι περιοχές υψηλού εισοδήματο. Αυτά λένε τα στατιστικά στοιχεία της ΦΑΟ. Χρησιμοποιούμε τα ίδια στοιχεία για, τον για τον πληθυσμό, για την παραγωγή, για το ΑΕΠ, την ίδια πηγή τη Στατιστική Υπηρεσία της ΦΑΟ. Αλλά στη μελέτη είναι, γίνεται πιο διεξοδική ανάλυση. Σε ό,τι αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στην ΚΑΠ, εκεί θα δίναμε έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς, συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό λέμε στη μελέτη, να στηρίξουμε με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις συγκεκριμένα προϊόντα που πραγματικά χρήζουν προστασίας και στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε από τις απορίες σας είναι το θέμα των μικρών καλλιεργητών και το θέμα της ε, εγκατάλειψης των ε, εκμεταλλεύσεων και των γεωργών. Όντως, αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Έχουμε τη γύρανση και του αγροτικού πληθυσμού και το γεγονός ότι οι νέες γενιές, οι νέοι, επιλέγουν άλλα επαγγέλματα. Αυτό είναι πρόβλημα. Επίσης, το φαινόμενο της αστιφιλίας. Το 70% ε, του πληθυσμού μέχρι το 2050 θα μένει σε αστικά κέντρα. Και αυτό όντω είναι μείζον ζήτημα. Αυτό το επισημάναμε. Τώρα, όταν εξετάζουμε τις επιλογές της πολιτικής, και εδώ δεν περιοριζόμαστε μόνο στο τέταρτο σενάριο, είναι πολλά και διάφορα τα σενάρια που το πραγματεύονται. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουμε, σε κανένα σενάριο δεν θα μπορέσουμε να θρέψουμε τον κόσμο αν δεν έχουμε γεωργού που θα παράγουν τρόφιμα. Οπότε θέλουμε δράσει να στηρίζουμε του νέου γεωργού και να πείθουμε του γεωργού να μην εγκαταλείπουν τη γεωργική δραστηριότητα. Αλλά έχουμε και τι υποδομέ, το ψηφιακό χάσμα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το 5G και τα θέματα του 5G. Αλλά δεν μιλούμε αρκετά για το ψηφιακό χάσμα μεταξύ τη υπαίθρου και των αστικών κέντρων. Έχουμε ολόκληρες περιοχές της Ευρώπης που δεν καλύπτονται από το διαδίκτυο. Δεν, υπάρχει, δεν έχει φτάσει εκεί η ψηφιοποίηση. Δεν υπάρχει προθυμία των παρόχων να καλύψουν και τις αγροτικές περιοχές παντού. Αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα και ε, είναι ένας από τους ε, παράγοντες για την απερίμωση της υπαίθρου. Μιλούμε τώρα για την ψηφιοποίηση, για τη νέα ε, αγορά και για την συνεργατική οικονομία. Αλλά αυτά ισχύουν μόνο όταν είναι κανεί εντό του ψηφιακού κόσμου. Αν είναι εκτό του ψηφιακού κόσμου, είναι εκτό και όλων των άλλων πλέον εκτιμάτων που αναφέραμε. Επίση, θα πρέπει να στηρίξουμε του μικροκαλλιεργητέ και επίση να αντιμετωπίσουμε τη γύρανση του αγροτικού πληθυσμού και να αποτρέψουμε την απερίμωση τη υπαίθρου, να μην εγκαταλείπουν οι γεωργοί τι καλλιέργειέ του. Σε ό,τι σενάριο και να επιλέξετε αυτά τα θέματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αντιμετωπίσετε. Άλλο ένα σχόλιο, ότι δεν ασχοληθήκαμε δεόντως με τη βιολογική γεωργία. Μιλούμε και για τη βιολογική γεωργία στη μελέτη. Είναι μια σημαντική τάση η βιολογική γεωργία και σίγουρα είναι μια τάση που ταυτόχρονα διασφαλίζει και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είναι σημαντικό θέμα η βιολογική γεωργία για την διόρθωση της κλιματικής αλλαγή. Αλλά το πρόβλημα της βιολογικής γεωργίας σήμερα είναι ότι υπάρχει μια σχετική συμβατότητα μεταξύ των βιολογικών προϊόντων σε ό,τι αφορά τις τιμές, είναι πιο ακριβά. Και έτσι είναι απρόσιτα τα προϊόντα αυτά σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού λόγω των ακριβών τιμών τους. Και όταν μιλούμε για την, το να ταΐσουμε τον πλανήτη, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Και ακόμη και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εντό Ευρώπη, έχουμε ομάδε πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγιεινά τρόφιμα. Εξού και το φαινόμενο της παχυσαρκίας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Και είναι σημαντικό να έχουμε βιολογικά προϊόντα, βιολογική γεωργία, αλλά για να πραγματικά θρέψουμε τον κόσμο, δεν αρκεί η βιολογική γεωργία, τουλάχιστον με τη σημερινή της μορφή, δεν αρκεί. Ούτε οι μικρές καλλιέργειες αρκούν. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία, από την ευρία έννοια, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης, ώστε να φέρουν τα βιολογικά προϊόντα και της μικρής ευέλειας γεωργία στο ευρύτερο τοπίο, στο, το, στο σενάριο. Γιατί αναφέρθηκατε στις πολυεθνικές ως απειλή για τους μικρούς καλλιεργητές. Γιατί θα μονοπολίσουν ε, και θα καταβροχθήσουν τους μικρούς καλλιεργητές. Αυτά και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ε, ε ευχαριστώ. Ήταν και δύσκολο να απαντήσει κανείς μέσα σε 10 λεπτά, σε λεπτομέρειες όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα θέλαμε όμως να τηρήσουμε και το πρόγραμμά μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, που παρουσιάσατε τη μελέτη και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει τους ερχόμενους μήνες όταν θα συζητήσουμε την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεν ήθελα να διακόψω εδώ τη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας μέχρι τις 2.30. Ε, ε, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. κυρία Μαγκίνη ζήτησε το λόγο. Συγγνώμη. Στα διάφορα έχω κάτι να πω. Υπάρχει ένα άρθρο του New York Times για τις πληρωμές της ΚΑΠ. Ε, θα το έχουν δει οι συνάδελφοι. Παρακαλώ να το δουν και οι συντονιστές. Γιατί δεν μας βοηθάει να υπερασπιστούμε τις δαπάνες της ΚΑΠ. Εάν ισχύουν όσα αναφέρει το διομοψίευμα αυτό το New York Times. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη αυτή. Μάλιστα, το διαβάσαμε κι εμείς. Δυόμιση ώρα συνεχίζουμε και σε πέντε λεπτά ε, τη συνεδρίαση των συντονιστών που δεν είναι δημόσια, όπως πάντα.